Συνάδελφοι, έχουμε πολύ γεμάτη μερίσια διάταξη απόψε, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Βλέπω την ομιλήτριά μας που ενημερώνεται για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ε, σήμερα το πρωί συμφωνήσαμε ότι θα εξετάζαμε το 14 πριν από το 13. Θα συζητήσουμε λοιπόν για μια μελέτη που ονομάζεται προ μια πιο αποτελεσματική παγκόσμια ανθρωπιστική δράση. Πώ μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη μελέτη τη ζήτησαν οι συντονιστές στην προεργασία για τη διάσκεψη κορυφή της Κωνσταντινούπολη την επόμενη χρονιά. Νομίζω, θέλετε, να, θέλετε να πείτε κάτι εισαγωγικά, όχι, ωραία, στη συνέχεια. Η μελέτη λοιπόν συντάχθηκε από το δικό μας ε, ε, τμήμα έρευνας. όχι, όχι, όχι, όχι αυτή η μελέτη, όχι. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχα τη συνεργασία. Μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι ήταν η κοινή μελέτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η μελέτη έχει εκπονηθεί από την κυρία Τσουράκα Μουγαρόσα από το Ισπανικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, καλωσορίσατε στην ε, συνεδρίασή μας. Ε, συζητήσαμε επανελειμμένως για τα τεράστια νούμερα εκτοπισμένων ανθρώπων, την αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να βρούμε χρήματα για να την αντιμετωπίσουμε. Σήμερα το πρωί στους συντονιστές μιλήσαμε για τα προβλήματα των παιδιών των προσφύγων, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αρκεί πλέον για να εγγυηθεί την εκπαίδευσή τους. Οπότε... Πολλά θέματα από αυτά θα είναι επιτάπητο στην επόμενη διάσκεψη αυτή κορυφή τη Κωνσταντινούπολη. Ποια είναι λοιπόν τα προβλήματα που υπάρχουν και τι θα πρέπει να ζητήσουμε να επιληθεί στη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, μέλη αυτής της Επιτροπής. Όπως είπε η κυρία Μακάβαν, Έχω όντως εργαστεί για αυτή την έκθεση που ανετέθη σε μας από την Επιτροπή σας. για το πώς θα, ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επόμενη διάσκεψη κορυφής για τα ανθρωπιστικά ε, ζητήματα. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν στο σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας, ποιοι θα είναι οι προσανατολισμοί της Ένωσης και διάφορα ε, οριζόντια θέματα Ποιε θα είναι κατάλληλε προτάσεις για το ρόλο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής. Ε, αν δεν είχατε την χρόνο ή την ευκαιρία να δείτε την έκθεσή μας, να σας πω ότι πρόκειται για μια επισκόπηση της, ε, των, πρω, των πρωτοβουλειών. Ποιες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες διαδικασίες διαβούλευσης που γίνονται φέτος Έχουμε μια θεματική απεικόνηση, επισκόπηση μάλλον των ε, βασικών θεμάτων. Είναι τα κεντρικά θέματα που έχουν συζητηθεί για την ανθρωπιστική δράση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η αποδοτικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας, δηλαδή ποια θα πρέπει να είναι η ανταπόκριση σύμφωνα με το πλαίσιο και ποιος είναι στην καταλληλότερη θέση για να ανταποκριθεί. Δεύτερον, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ευάλωτο χαρακτήρα ε, και πώς θα μετακινηθούμε από τη διαχείριση κινδύνου μάλλον από την ε, άμεση ανταπόκριση σε καταστροφές ε, στην διαχείριση του κινδύνου, πώς ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες σύγκρουσης και πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην ανθρωπιστική μας δράση, δηλαδή μετατροπές και ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες. Αυτές είναι οι βασικές προκλήσεις και έπειτα κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσαρμοσμένη σε όλα αυτά και κάποιες συστάσεις. Ήθελα να σας αναφέρω ποια πιστεύω ότι είναι τα βασικότερα ζητήματα. Καταρχήν, γιατί διοργανώθηκε η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την ανθρωπιστική βοήθεια. Καταρχήν ήταν μια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και αναφέρει την ιδέα της προσαρμογής του ανθρωπιστικού συστήματος και της ανθρωπιστικής δράσης και ζήτησε να διοργανωθεί μια διάσκεψη κορυφής για την ανθρωπιστική δράση. Γιατί? Γιατί έγιναν συζητήσεις σε πολύ σημαντικές μετά από την ανταπόκριση στην ΑΙΤ, στο τσουνάμι και τέθη το ερώτημα πώς θα ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες, το αυξανόμενο κόστος της βοήθειας, τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πιο παρατεταμένες κρίσεις. Υπάρχουν εμπόδια ε, από πλευράς ανθρώπινων πόρων αλλά και οικονομικών πόρων και πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις παγκόσμιες τάσεις που δείχνουν ότι θα υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στο μέλλον, όπως η έλλειψη του νερού, τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών και ούτω καθεξής. Πώς λοιπόν μπορούμε να ανταποκριθούμε και πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε τις τοπικές και εθνικές ε, προσπάθειες ώστε να σκεφτούμε με νέο τρόπο και να μπορέσουμε να ενεργήσουμε μέσα στα, στους περιορισμούς του συστήματος. Ο στόχος είναι να συμφωνηθεί μια, ένα θεματολόγιο από το 2016 και έπειτα που θα είναι πιο ολοκληρωμένο, θα λαμβάνει υπόψη τους διάφορους φορείς και να είναι ε, ε, ε, κατάλληλο ώστε να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές ανάγκες. Ε, θεωρείται μια ιστορική σημασία σε ευκαιρία γιατί ε, συνδέεται με την χρηματοδότηση της ανάπτυξης, με τη διάσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές και Υπάρχει μια έκθεση για την οικοδόμηση της ειρήνης και τη διατήρηση της ειρήνης και στις 21 Μαΐου ο Μπάν Κιμούν δημιούργησε ένα πάνελ ε, ψηλού επίπεδου για την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε λοιπόν ε, κάποιους άξονες για διαβουλεύσεις. Έχουμε 8 περιφερειακούς άξονες ε, και μία παγκόσμια διαβούλευση. Υπάρχουν διάφορες θεματικές διαβουλεύσεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται ε, online διαβούλευση όπου οποιοδήποτε μπορεί να παρέμβει στο διαδίκτυο και στο site της ε, ε, Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Ανθρωπιστική Δράση και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά σε αυτή τη διαφάνεια, πάντως αν τη βλέπετε βλέπουμε τις διάφορες θεματικές διαβουλεύσεις που τρέχουν, ενώ ταυτόχρονα γίνονται και online διαβουλεύσεις και έχουμε και θεματικές ομάδες. Είναι μια ευρύτατη λοιπόν διαδικασία με την ιδέα να είναι ολοκληρωμένα, είναι περιστατωμένη. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά οι ΜΚΟ, οι διεθνείς οργανισμοί, οι κοινότητες που έχουν πληγεί, οι κοινότητες της διασποράς, ο πανεπιστημιακός κόσμος και ο ιδιωτικό τομέας βεβαίως. Ποια είναι τα τέσσερα βασικά θέματα τι πρέπει δηλαδή να αλλάξει στο σύστημα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πώς θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, πώς θα μειωθεί ο κίνδυνος, πώς θα βοηθήσουμε εκείνους που επηρεάζονται από συγκρούσεις και έπειτα πώς θα γίνει πιο αποδετική η διαχείριση και πώς θα επιταχυνθούν οι αλλαγές. Διάφορες προτεραιότητες έχουν ήδη προκύψει από τις διαβουλεύσεις. Η πρώτη που υπογραμμίζεται σε όλες τις διαβουλεύσεις είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της απάντησης που θα δοθεί. Η προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στους πιο ευάλωτους και επίσης η σημασία της χειραφέτησης των, πληθυσμών, ε, των πληγέντων πληθυσμών, κυρίως των γυναικών, αλλά και λογοδοσία αφοσίωση και σεβασμός των ανθρωπιστικών αρχών και του διεθνούς νομικού πλαισίου. Ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια είναι η πρόσβαση στους πληθυσμούς. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε για παγκόσμιες στάσεις που επηρεάζουν το μέλλον της ανθρωπιστικής δράσης. Το 80% της χρηματοδότησης φαίνεται να πηγαίνει στους πληγέντες λαούς και έχουμε ως προτεραιότητες στη Συρία, τον Νότιο Σουδάν και το Ιράκ. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα λοιπόν στην ε, ανθρωπιστική δράση και στην προστασία που δίδεται μέσω αυτής. Επίσης θα πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα συστήματα στα εθνικές και περιφερειακές ανάγκες. Ένα άλλο κεντρικό θέμα είναι η αλλαγή του, του παραδείγματος, δηλαδή των υποθέσεων που κάνουμε, να μπορέσουμε να προβλέψουμε και έτσι αυτό πρέπει να το συνδέσουμε και με τις συζητήσεις περί αναπτυξιακής βοήθειας. Βασικές εταιρικές ε, σχέσεις, συνεργασίες, ε, όχι μόνο με τις ΜΚΟ, τον ιδιωτικό τομέα, τον, τους πανεπιστημιακούς, όλοι μαζί θα πρέπει να σκεφτούμε νέους τρόπους για να ανταποκριθούμε και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις και όρους για καινοτομία. Είναι διάφορα θέματα λοιπόν, προσπάθησα να σας τα συνοψίσω ε, για τα τέσσερα αυτά ζητήματα υπάρχουν και διάφορα κάθετα θέματα που διαπερνούν όλους τους τομείς. Έχουμε ανάγκες, ε, μάλλον έχουμε, θέλουμε να έχουμε προσεγγίσεις που βασίζονται στις ανάγκες και στο πλαίσιο, αλλά που θα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και στα διαφορετικά πλαίσια. Έπειτα, η ε, δυνατότητα να επηρεάσουμε τον κόσμο και της κοινότητας να εντοπίσουμε τις απαντήσεις μας, η έγκαιρη, ευέλικτη και προβλέψιμη χρηματοδότηση, αλλά και το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε άλλες περιστάσεις, όπως ας πούμε σε αστικά πλαίσια, γιατί ο πόλεμος ας πούμε στη Συρία τώρα γίνεται στις ε, πόλεις και σε χώρες μεσαίου εισοδήματος, καθώς και η ανάγκη να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τις εταιρικέ σχέσεις στο ανθρωπιστικό σύστημα. Τώρα, τρία βασικά αιτήματα φαίνεται να προκύπτουν από τις διάφορες περιφέρειες. Η ανάγκη να προστατευθούν και να, οι λαοί αλλά και να τους δοθεί αξιοπρέπεια να βρούμε καινοτόμε και βιώσιμες λύσεις, αλλά και να εντοπίσουμε σε συγκεκριμένα σημεία την ανθρωπιστική ανταπόκριση. Το να τοποθετηθεί η προστασία στο επίκεντρο. Αυτό είναι μια κραυγή που προκύπτει από τις περισσότερε περιφερειακές διαβουλεύσει. Η προστασία είναι το κυριότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Συζητάμε πολύ το θέμα των φυσικών καταστροφών, των κλιματικών αλλαγών, Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα του πώς θα προστατέψουμε τον κόσμο που επηρεάζεται από τη βία. Δηλαδή, ε, αντί να αντιδρούμε θα πρέπει να μπορέσουμε να προλάβουμε. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Κάτι ακόμα είναι το πώς η ανθρωπιστική δράση θα αποτελέσει τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ώστε να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα της σύγκρουσης χωρίς αυτό να εμποδίσει τις ανθρωπιστικές δράσεις. Βλέπουμε τώρα διάφορες εντάσεις Ε, γιατί υπάρχει και το θέμα του πού σταματάει η ανθρωπιστική δράση. Είναι μόνο μια γρήγορη ανταπόκριση, μια γρήγορη απάντηση ή πηγαίνει και στην αποκατάσταση και στην ανάπτυξη. Εξαρτάται κάθε φορά και από το πλαίσιο. Η ανησυχία ότι εν τέλει η ανθρωπιστική δράση είναι η απάντηση σε μια αποτυχία της ανάπτυξης και της ε, ανικανότητας να ληφθούν πολιτικές ε, αποφάσεις και άρα η ανησυχία είναι ότι φαίνεται η ανθρωπιστική δράση να είναι ε, η απάντηση, αλλά δεν είναι η απάντηση. Είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όταν η ανάπτυξη και οι πολιτικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί όταν έπρεπε. Οι εντάσεις που εμφανίζονται σε πολλές χώρες ε, επηρεάζουν την εξωτερική ανθρωπιστική δράση. Για παράδειγμα, έχουμε την κατάσταση στη Συρία. Το Συριακό κράτος προσπαθεί να αποποιηθεί τον ευθυνών του, να αποφύγει τις ευθύνες. Και μερικές φορές ε, οι χώρες, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θέλουν να ληφθούν, θέλουν να, να λαμβάνουν την υπόψη και δική τους θέση. Θα μείνει πόσο δεκτικές είναι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Και το θέμα δεν είναι ε, ε, μόνο το θέμα της ε, πώς γίνεται αντιληπτή η ανθρωπιστική δράση, γιατί πολλές χώρες όπως οι Ισλαμικές δεν, δεν ακολουθούν την αρχή της ανθρωπιστικής δράσης, αλλά στηρίζουν την ανθρωπιστική δράση στην αλληλεγγύη, αλλά δεν σκέφτονται με τέτοιες αρχές. Ποιες είναι οι βασικές τώρα προκλήσεις Καταρχήν η διαδικασία είναι μία πρόκληση. Γιατί είναι μία ευρύτατη διαδικασία και πολλοί λαμβάνουν μέρος, πολλοί φορείς. Αλλά φαίνεται να είναι ανοιχτή η διαδικασία, ατέρμονη. Και η βασική πρόκληση είναι ότι το θεματολόγιο ακολουθεί μία θεματική κατανομή. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει θεματολόγιο, αλλά εκεί αποφασίζονται τα βασικά προβλήματα που ανακύπτουν από τις διαβουλεύσεις. Και μερικοί πιστεύουν και επικρίνουν την έλλειψη διαφάνειας ή τουλάχιστον επαρκούς διαφάνειας στην όλη διαδικασία. Δεν μου έχει απομείνει και πολλούς χρόνους και αυτό θα περάσω στο θέμα της ε, ευρωπαϊκής ε, συνεισφοράς στην ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω ε, ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε με, το, με αυτό που κάνουμε καλύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να συμβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο και πού διαφέρουμε σε σχέση με άλλους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, εδώ μιλώ για την ΕΚΟ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το ΕΚΟ. Το ΕΚΟ είναι από τους μεγαλύτερους δωρητές, αλλά όχι μόνο. Το γραφείο ΕΚΟ θεωρείται ότι προωθεί και τις βέλτιστες πρακτικές μέσω της ε, Ευρωπαϊκής Συνένεσης και θεωρείται πραγματικά δωρητής με βάση την ε, αρχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι λοιπόν χρήσιμη και η ανθρωπιστική αρχή και η Ευρωπαϊκή Συνένεση και αυτά θα μπορούσαν να περιληφθούν στη διακήρυξη της διάσκεψης κορυφής για την ανθρωπιστική βοήθεια ως υποδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και έχει προσαρμοστεί στην κατάσταση προκειμένου να αντιδρά με καλύτερο τρόπο και με επάρκεια ανάλογα με την ανάλυση του κινδύνου, ανάλυση του ευρύτερου πλαισίου και το ΕΚΟ έχει πραγματικά μια μοναδική θέση ως περιφερειακός δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί ως περιφερειακή οργάνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μοναδικότητα και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γραφείου της για την ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί βλέπουμε όλο και πιο τροτές χώρες, όλο και πιο ευάλωτες. Βλέπετε την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ, το πρόβλημα με το Ισλαμικό κράτος. Εκεί χρειαζόμαστε όλο και περισσότερες περιφερειακές οργανώσεις κατά το πρότυπο του ΕΚΟ, του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το ΕΚΟ, χάρη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατάφερε να έχει επαρκή και ε, επίκαιρη χρηματοδότηση για να αποφευθούν κενά στη χρηματοδότηση. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ ανέκαθε θεωρούσε τους πληγέντες πληθυσμούς ε, ως βασικούς δικαιούχους της ανθρωπιστικής βοήθειας και προσπαθούν ε, ώστε να μην χρησιμοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια ως πολιτικό ε, μέσο ή εργαλείο και συνεργασία με τους εταίρους είναι κάτι που επίσης ενδιαφέρει την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Κάτι άλλο που προωθεί το γραφείο ΕΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία της αντοχής, η δημιουργία θεκτικότητας και μείωση της, του κινδύνου καταστροφής. Και εδώ υπάρχει συνεργασία και με άλλους διεθνείς δωρητές. Και σε ό,τι αφορά την καινοτομία, για πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια το ΕΚΟ προωθεί έναν καινοτόμο τρόπο προβολής προγραμμάτων σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, έρχομαι προς το τέλος και τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να προωθηθεί η Ευρωπαϊκή Συνένεση ως πρότυπο για την Παγκόσμια Συνένεση για την Ανθρωπιστική Δράση. Και ένα από τα βασικά θέματα τα βασικά προβλήματα ότι δεν υπάρχει συμφωνία για την αρχή της ανθρωπιστικής δράσης. Γι' αυτό και χρειάζεται ένα παγκόσμιο σύμφωνο και μακάρι αυτό να είναι το αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής της Κωνσταντινούπολης. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να στηρίξουν και να προωθήσουν αυτή την Ευρωπαϊκή Συνένεση και την Παγκόσμια Συνένεση και να πρωτοστατήσουν στην διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της διάσκεψης κορυφής. Αυτή τη στιγμή η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και κάποιες χώρες μέλη είναι πολύ διακριτικές και κρατούν στάσεις σιωπής. Απλώς ακούν και αφουγκράζονται τις εξελίξεις, αλλά εν ώψη και της επικείμενης διάσκεψης κορυφής, τώρα είναι η στιγμή για να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να καθοδηγήσει για να χαράξει το δρόμο προς την Κωνσταντινούπολη, πρωτοστατώντας τις εργασίες. Επίσης, θα πρέπει να συνδέσουμε ε, τη διαδικασία αυτή με το πλαίσιο μετά την, ε, την, το αναπτυξιακό θεματολόγιο και το τι θα γίνει μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Μου λέτε ότι πρέπει να ολοκληρώσω. Μάλιστα. Προστασία, η προστασία θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής. Κάτι που κάνει ήδη το ΕΚΟ. Αλλά πολύ περισσότερο από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό ζητούν και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αυτό προέκυψε και από τι διαβουλεύσεις και επίση θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό συμβούλιο για τα ανθρωπιστικά θέματα. Ένα ειδικό Υπουργικό Συμβούλιο που θα ασχολείται μόνο με τα ανθρωπιστικά. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ε, τάση να εντάσσεται η ανθρωπιστική δράση στι υπόλοιπε εξωτερικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ καλό θα ήταν να τη δίνεται ξεχωριστή σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι ένα υπόδειγμα περιφερειακής διαδικασίας ολοκλήρωσης και είναι η μοναδική οργάνωση στον κόσμο που έχει την ικανότητα και τα μέσα, τα εφόδια να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αίτια του κακού, τα αίτια των κρίσεων και των συγκρούσεων. Έτσι, ο συνδυασμός με τη μείωση της ε, του κινδύνου καταστροφών αλλά και την παροχή ανθρωπιστικής αρρωγής είναι σημαντικό. Δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε όμως την ανθρωπιστική ε, απάντηση με τις άλλες εξωτερικές πολιτικές γιατί έτσι ε, αλλοιώνεται κάπως το περιεχόμενό της. Λυπούμε που χρειάστηκε να μιλήσω με μεγάλη ταχύτητα γιατί είχα αλλάξει το χρόνο, ζητώ εκ των υστέρων συγγνώμη από τους διερμηνείς σε που δεν κατάφεραν να με παρακολουθήσουν. 20 λεπτά μιλήσατε ενώ είχατε 10 στη διάθεσή σας. Ωραία, τώρα λοιπόν, ε, ποιοι παρακαλώ θα ήθελαν ε, το λόγο. Έρικ, βέβαια εσύ, ε, θα, βέβαια, έχεις χρόνο. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το οποίο δυσκολεύομαι να καταλάβω για την ανθρωπιστική δουλειά της Κομισιόν και το κείμενό σας, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι κάναμε λάθος στην ΑΕΤ που πρέπει να διορθώσουμε, ποια προβλήματα πολιτικής, γιατί έχουμε αυτή τη συνάντηση γιατί θέλουμε να συμμετάσχουν και άλλοι στην προσπάθεια, γιατί κάποιες χώρες ε, θα βοηθήσουν με χρηματοδοτήσεις. Ποια είναι τα πραγματικά πολιτικά θέματα. Ξέρουμε ποια είναι τα θέματα. Έτσι θα μάθουμε καλύτερα ποια είναι τα θέματα. Αν θέλουμε απλώς να πούμε ε, ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός για όλους, όλα αυτά μοιάζουν ε, λίγο ευχολόγιο. Τι είναι ακριβώς το πλαίσιο. Αλλά Ερικ, ε, που είσαι ο εισηγητής μας. Ο Ενρίκε, α, ο Ενρίκε Γερέρο, που είναι ο εισηγητής μας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ, Χριστίνα, ευχαριστώ για την εργασία που επετέλεσες και για το τι έκανε την παρουσία σου στα αγγλικά, γιατί αν δεν είχε κάνει στα βάσκικα θα είχαμε σοβαρές δυσχέρειες κατανόησης. Ξέρω τι εργασία έχεις κάνει για να εκπονήσεις ένα τέτοιο κείμενο που έχει βέβαια λίγες σελίδε, αλλά για να καταλήξεις αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να κάνεις πολλή δουλειά. Και αυτό που πραγματικά σε εμπνέει δεν είναι βέβαια η αμοιβή που θα λάβεις, αλλά το ότι θα βοηθήσεις τη διαμόρφωση της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη της συνάντησης κορυφής για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη του χρόνου και πώς θα επιχειρήσει να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα είναι ο εκπρόσωπος ε, των θέσεων της Ένωσης. Δέχομαι την πρόκληση στην οποία αναφέρθηκε η Λίντα όταν είπε τι θέλουμε να επιτύχουμε με αυτήν την ανθρωπιστική συνάντηση κορυφής. Έχει πολλούς λόγους για τους οποίους το διοργανώσαμε. Αλλά ο κύριος είναι ότι πρέπει να ξαναδούμε το θέμα σε διάφορους τομείς μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα διότι από το 1991 που τα Ηνωμένα Έθνη ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα ο κόσμος έχει αλλάξει από πολλές πλευρές ε, ορισμένες είναι λόγω φυσικών λόγων αλλά και λόγω της παρέμβασης του ανθρώπου έχουμε τώρα περισσότερες κρίσεις που προκαλεί ο άνθρωπος ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε τόσες ανθρωπογενείς κρίσεις σε ένα επίπεδο που Φύγονται πολύ περισσότεροι, πρέπει να ανταποκριθούμε με περισσότερες πιστώσεις. Αλλά πάνω απ' όλα αντιμετωπίζουμε κρίσεις που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, αλλά επίσης από νέους που παρεμβαίνουν, νέους παράγοντες που παρεμβαίνουν ε, στη διεθνή σκηνή, νέες αναδιόμενες χώρες, αλλά και άλλες χώρες που επίσης προσπαθούν να τοποθετηθούν για να παίξουν ρόλο στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια, στην αντίδραση στα ανθρωπιστικά προβλήματα, διότι έχει αναπτυχθεί πολύ περισσότερο η κοινωνία των πολιτών, υπάρχει ένα δίκτυο μη κάπα όμικρον πολύ πιο εκτεταμένο, υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για διάφορα θέματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση. Απαντώ απευθείας πολύ απευθεία στην ερώτηση της Λίντα. Μπορώ να πω ότι με τον ίδιο τρόπο που τα Ηνωμένα Έθνη στην αρχή του, της χιλιετίας υιοθέτησε τους στόχους της ε, χιλιετίας για να εντοπίσει ελλείμματα στην εκπαίδευση, στη φτώχεια, την υγεία, την ε, παιδική θνησιμότητα, την κατάσταση των γυναικών κλπ. κλπ. Με τον ίδιο τρόπο η διεθνής κοινότητα χρειάζεται επίσης να ξαναδεί τη γενική της πολιτική αντίδρασης τι ανθρωπιστικές κρίσεις. Αυτός είναι ο θεμελιώδης στόχο της συνάντηση Κορυφή που έχουν συγκαλέσει τα Ηνωμένα Έθνη του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, Εντό τη διαδικασίας προς αυτή τη συνάντηση κορυφή, πρέπει να δούμε τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ένωση. Όχι μόνο ότι έχει αλλάξει στη σκηνή συνολικά, την παγκόσμια, αλλά και ποιες είναι οι προτεραιότητες που εμείς ως ε, φορείς της ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούμε να κάνουμε για να επιτύχουμε συνένεση γύρω από τους στόχους αυτούς σε αυτή τη συνάντηση του χρόνου. Τις αλλαγές στην παγκοσμία σκηνή ε, την ανέφερες, τις ανέφερες, αλλαγή αυτών που παρεμβαίνουν, αλλαγή στα αίτια της κρίσης, έλλειμμα χρηματοδότησης, Πολύ διαφορετική κατάσταση στον κόσμο. Τώρα για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πω αργότερα. Ποιες είναι τώρα οι προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα. Καμιά φορά διαρωτώμεθα ποιος είναι ο βασικός στόχος ανθρωπιστικής βοήθειας. Να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των θυγωμένων. Που υποφέρουν από μια θεομηνία ή λόγω των επιπτώσεων μια κρίση που προκλήθηκε από μια πολιτική σύγκρουση. Να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες αυτές, να τα αποκριθούμε. Δηλαδή, από ανθρωπιστική άποψη, να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες χωρίς να έχουμε καμία πολιτική σκοπιμότητα. Να λάβουμε υπόψη δηλαδή ότι οι αρχές της ανθρωπιστική δράσης είναι η ανεξαρτησία, η ουδετερότητα κτλ. Οι αρχέ αυτέ πρέπει να είναι χαρακτηριστικά της αντίδρασης μας. Είμαστε εκεί για να σώσουμε ζωές. Είναι αυτοί που είναι εκεί επί τόπου ενώ βεβαίω. Όχι εγώ ίδιος βεβαίως, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί που είναι εκεί επί που διευθύνουν τις οργανώσεις που χορηγούν την βοήθεια αυτή για να αντιμετωπιστούν απευθείας τα προβλήματα, να σωθούν ζωές, να τους χορηγήσουμε τα βασικά αγαθά επιβίωσης, ε, για να τους χορηγήσουμε εκπαίδευση στα παιδιά, να τους δώσουμε γιατρική περίθαλψη. Πριν τεθεί οποιοδήποτε άλλο θέμα για ποια είναι η χρησιμότητα, ποιες είναι οι πολιτικές ε, επιλογές κτλ. Αυτή η αρχή in but out. Ναι μεν βοηθάμε αλλά κρατάμε και την απόστασή μας. δεν είναι τμήμα πολιτικών ε, στρατηγικών για την επίλυση των κρίσεων. Αυτό θέλουμε να πούμε. Αυτό είναι ορισμένε φορέ δύσκολο να το προβάλλει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί διατρέχουμε τον κίνδυνο φυσικά να συμμετάσχουμε στη γενικότερη στρατηγική παρουσία της Ένωσης ε, στον κόσμο, δηλαδή να υποταχθούμε στην πολιτική ανάπτυξη. Ενώ εμάς ο στόχος μας είναι η άμεση αντίδραση στις ανάγκες και κατόπιν στη δημιουργία μιας σύνδεσης μεταξύ αυτών των αναγκών και μιας πολιτικής ε, ανάρτησης πιο ουσιώδους. Γιατί ξέρουμε ότι πολλές ε, κρίσεις παρατείνονται, κρατάνε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται μόνο άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Δεύτερον, δεύτερον μια προληπτική προσπάθεια και της χορήγησης ε, δυνατοτήτων στον τοπικό πληθυσμό σε πολλές περιπτώσεις κρίσης, αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε ούτω ώστε να έχουν οικονομική διακυβέρνηση και πολιτική διακυβέρνηση μέσω άλλων μη ανθρωπιστικών πολιτικών, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τις ε, συγκρούσεις αυτές. Αλλά είναι σαφές, όπως απεδείχθηκε και στην ε, συνάντηση κορυφής πρόληψης κινδύνων στο ΣΕΝΤΑΙ, ότι η καλύτερη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε θεομηνίες είναι η εκπαίδευση των πολιτών, η χορήγηση δυνατοτήτων, να βοηθήσουμε δηλαδή, να δώσουμε περισσότερες δυνατότητε στις ε, τοπικές αρχές, στις εθνικές αρχές, στην κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις που δρούν επί τόπου. Τρίτη προτεραιότητα, να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους. Στις ανθρωπιστικές κρίσεις, οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, αυτοί αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πρέπει να έχουμε πολύ συγκεκριμένα προγράμματα για να βοηθήσουμε τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Υπόθηκε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ της άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας με την ανάπτυξη όταν οι κρίσεις αυτές παρατείνονται. Μηχανισμοί χρηματοδότησης. Έχουμε δει τελευταία τι έγινε με το πρόγραμμα των Ηνωμένων ε, Εθνών ε, για τα τρόφιμα που χρειάστηκε να ανασταλεί στην περίπτωση της, χειρίας, στις Συρίας διότι δεν υπήρχαν πιστώσεις. Πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια εξέβρεσης νέων πόρων να εμπλακούν δηλαδή και άλλοι σε αυτήν την ε, ανθρωπιστική αντίδραση. Επίσης αναφέρθηκες στο ρόλο που πρέπει να παίξει η κοινωνία των πολιτών και στην ενίσχυση των κυβερνήσεων των αρχών σε διάφορα επίπεδα και αναφέρω, τονίζω αυτό που είπες, ότι πρέπει να προστατεύουμε και αυτούς που δρούν επί τόπου. Ο αριθμός του προσωπικού χωρίς ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει πεθάνει, που έχει σκοτωθεί σε περιοχές όπου έχουμε συγκρούσεις, αυξάνεται και νομίζω ότι οι διάφορες κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανώσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Τρίτο και προχωρώ. Ρόλος της Ένωσης. Εν ώψη της ε, συνάντησης κορυφής, αλλά και μετά. Εν ώψη της συνάντησης κορυφής. Ξέρουμε επιτέλους ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια ανακοίνωση τον προσεχή Σεπτέμβριο. Έχουμε ήδη ε, κάποιες ε, ιδέες για το ποιες θα είναι οι βασικές γραμμές που σχετίζεται και με την εργασία που εσύ επετέλεσες και, σε, και σχετίζεται και με αυτά που είπε η Επιτροπή μας επί του θέματος αυτού. Το Συμβούλιο από την πλευρά του. Αν και, αν και, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, η συνάντηση κορυφής αυτή δεν θα είναι διακυβερνητική. Δεν θα είναι όπως οι άλλες τέτοιες συναντήσεις κορυφής που έχουν γίνει φέτος όπου διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνήσεις συμμετέχουν ως εκπρόσωποι σε αυτές τις συναντήσεις κορυφής. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν το ρόλο της Ένωσης εκφράζοντας σαφώς ως Συμβούλιο μια άποψη. Γιατί το Συμβούλιο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ξέρουμε ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου ενδιαφέρεται πολύ για αυτή τη συνάντηση κορυφή και η Ολλανδία που είναι η μετέπειτα Προεδρία. Θα θέλαμε λοιπόν μια απόφαση του Συμβουλίου τον Οκτώβριο, νομίζω ότι αυτό προβλέπεται, αν θυμάμαι καλά, για να τονίζει ότι έχει ρόλο σημαντικό η Ένωση με τη συμμετοχή των κρατών μελών, αν και δεν θα είναι σύνεδροι λοιπόν σε αυτήν την συνάντηση κορυφής. Και όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο θα προετοιμάσει μια έκθεση πρωτοβουλίας της οποίας εγώ θα είμαι ο εισηγητής. Και χάρη στην ε, Αναρίκα έχουμε ένα πρώτο σχέδιο που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Ανάπτυξης αρχές Οκτωβρίου. Επίσης, επίσης Και θυμάμαι και αυτό που είπε ο Ντάβορ. Έχουμε τη δυνατότητα στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι μπορούμε να πιέσουμε ούτω ώστε να υπάρξει επαρκής αναφορά σε αυτές τις δύο συναντήσεις κορυφής στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων. Και ο άλλος ρόλος που πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κωνσταντινούπολη είναι η πείρα τη, οι βέλτιστες πρακτικές και η κοινή πεποίθηση ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής μας. ούτω ώστε να υπάρξει μια παγκόσμια συνένεση για το ότι πρέπει να είναι παγκόσμια προτεραιότητα. Και κατά λίγο μετά την Κωνσταντινούπολη τι πρέπει να κάνουμε. να δούμε και να συζητήσουμε εδώ ως Επιτροπή εάν θα αναθεωρήσουμε τον κανονισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης με βάση και τις δεσμεύσεις και συμφωνίες που θα έχουν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή πώς θα διαμορφώσουμε τη δράση μας στον τομέα αυτό για τα επόμενα 10-15 έτη. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να προβλέψουμε τη δημιουργία ενός παγκοσμίου ταμείου ανθρωπιστικής βοήθειας με εθελοντικές αλλά και υποχρεωτικές συνεισφορές. Οι υποχρεωτικές θα είναι για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις επέδου 3 και αυτές που θα προκύψουν ε, ευνίδια όπως ε, η κρίση έμπολα. Θα πρέπει δηλαδή τα κράτη-μέλη να προβλέπουν στους προπολογισμού τους κονδύλια για την ανθρωπιστική βοήθεια και θα το έχουμε υπόψη και όταν θα γίνει αναθεώρηση των πολιτών προοπτικών, πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών για να προσέξουμε να συμπεριλάβουμε και εκεί τα αναγκαία κονδύλια και η Επιτροπή μας έμαθε σήμερα το πρωί ότι λήφθηκε μια απόφαση για να θέσουμε το θέμα της εκπαίδευσης να έχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ούτω ώστε στα πλαίσια της αντιμετώπισης των, των ανθρωπιστικών κρίσεων να φροντίσουμε για την ανάπτυξη των παιδιών που είναι τόσο ευάλωτη ομάδα και που αν δεν εκπαιδευτούν όσο είναι παιδιά θα αντιμετωπίζουν ένα μειονέκτημα στην υπόλοιπη ζωή τους. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Ε, ξέρω, ξέρετε ότι είμαι αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Πολύ συχνά δίνω το λόγο, προβλέπω λίγο χρόνο ομιλίας και μετά όταν εγώ έχω τη δυνατότητα να μιλήσω, μιλάω περισσότερο από τους υπόλοιπους οποίους έχω δώσει το λόγο. Οπότε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και συνάδελφοι έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Απλά σας το λέω γιατί έχουμε τρία ακόμα θέματα με προσκεκλημένους ομιλητές. Πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα. Θα έχουμε όμως χρόνο και στο μέλλον. Γι' αυτό θα ήθελα να περιοριστείτε στο δίλεπτο αν είναι δυνατόν. Να το έχουμε κλείσει μέχρι τις 4 γιατί μετά έχουμε το φύλλο, μετά έχουμε τη Δυτική Αφρική και κάθε ένα από τα θέματα θα μας πάρει μια ώρα. Χέιντι. Ευχαριστώ. Ε, εντάξει, τότε δεν θα κάνω σχόλια. Έχω ένα σημείο, ένα λεπτό. Και είναι το εξή. Πώς λαμβάνετε υπόψη η κατάσταση των όσων ζουν στα, στα τόπεδα προσφύγων. Και αυτό το ρωτώ γιατί βλέπω συχνά πως οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα στρατόπεδα που μετατρέπονται σε μικρές πόλεις τελικά δεν έχουν καμία προοπτική για τη ζωή μετά από το στρατόπεδο ακόμα και αν ζήσουν εκεί για 20 χρόνια, όπως οι Σομαλοί στα, στα τόπεδα της Κένιας. Σε αυτήν την διάσκεψη θα εξεταστεί το θέμα των στρατοπέδων προσφύγων. Υπάρχουν καινοτόμε προσεγγίσεις για το πώς θα βελτιωθούν αυτά τα στρατόπεδα για να προετοιμάζουν τον κόσμο ώστε να επιστρέψουν στην φυσιολογική ζωή. Ευχαριστώ, Χέντι, που ήσουν και τόσο σύντιμη. Πάβελ. Ευχαριστώ, Λίντα. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση και για την παρουσίαση, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για την διάσκεψη κορυφής. Σε μια από τις διαφάνειες, στην προηγούμενη, υπήρχε μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την οποία θέλω να σας ρωτήσω. Γράψατε να στηριχτεί η δημιουργία ενός ειδικού σχηματισμού του Συμβουλίου για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, ώστε να μην υπάρχει ε, σύγχυση ανάμεσα στην ανθρωπιστική δράση της Ένωσης και την εξωτερική της πολιτική. Υπάρχει το Συμβούλιο των Υπουργών Ανάπτυξης που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και για τα αναπτυξιακά θέματα και τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Τι εννοείται με αυτή τη φράση, πρέπει αυτό να χωριστεί αφού η αναπτυξιακή πολιτική και τα ανθρωπιστικά ζητήματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση και μετά θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Η ερώτησή μου είναι η ίδια, γιατί είπατε στο τέλος σύντομα ότι δεν πρέπει να συγχαίεται η εξωτερική πολιτική με την ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα, ας είμαστε ειλικρινείς. Αν δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, δεν μπορούμε να μιλάμε πάντα με διπλωματικό λόγο, να πούμε ποιο είναι το πρόβλημα ξεκάθαρα και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Και αυτό που είπες ότι δεν είναι διακυβερνητική ε, διάσκεψη, ίσως εσύ θα μπορούσες να μας εξηγήσει, αλλιώς η κυρία Τσουχόκα. Να δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν γιατί δεν έχει ζητήσει άλλος συνάδελφος το λόγο. Uh, Κουάσι επίσης και κύριο Στράιτεν. Παρακαλώ σύντομα. Απαντήστε στα βασικά θέματα. Όχι, δεν έχουμε προετοιμασμένη ομιλία. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της έκθεσης. Απλά θέλω να επαναλάβω ότι θα γίνει ε, ανακοίνωση το Σεπτέμβριο με στρατηγική, ε, μας, το στρατηγικό μας όραμα το καλοκαίρι. Θέλουμε να εστιάσουμε στα θέματα μέσω μιας συλλογική ε, προσέγγισης να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς θα είναι πιο αποτελεσματική και αποδοτική ανθρωπιστική δράση. Ελπίζω λοιπόν ότι τις απαντήσεις θα τις βρείτε μέσα σε αυτή την ανακοίνωση και μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα συνεργαστούμε και με ορισμένους από τους εκπροσώπους εκπροσώπους το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Οι ε, καλεσμένοι μας τώρα. Ευχαριστώ για τους πρόσφυγες ή όσους διαμένουν σε καταβλισμούς προσφύγων. Το βασικό θέμα δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τι γίνεται με πρόσφυγες που δεν βρίσκονται σε καταβλισμούς. Γιατί για πολλά χρόνια η πραγματικότητα έχει δείξει ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες βρίσκονται εκτός καταβλισμών προσφύγων. Μένουν ε, σε πόλεις και το θέμα είναι τις δικές σου ανάγκες πώς θα τις καλύψουμε. Το πρόβλημα με τους καταβλισμούς προσφύγων είναι ότι έχουμε κάποιες εθνικές κυβερνήσεις που αποφασίζουν αν μπορούν να παραμείνουν ε, ή να, θα πρέπει να φύγουν από τους καταβλισμού οι πρόσφυγες. Και αυτές το αποφασίζουν. Πάντω ε, η βασική συζήτηση στη διάσκεψη κορυφής για τα ανθρωπιστικά θέματα είναι πώ θα καλυφθούν οι ανάγκε των προσφύγων που βρίσκονται σε διέλευση, διαμετακόμιση, βρίσκονται εκτός των καταβλισμών, γιατί οι περισσότεροι βρίσκονται εκτός καταβλισμών. Τέθηκε μία ερώτηση γιατί πρότεινα ξεχωριστό Συμβούλιο Υπουργών ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια διαφορετικό από αυτό της εξωτερικής πολιτικής. Παρόλο που υπάρχει διασύνδεση εξωτερικής δράσης και ανθρωπιστικής πολιτικής. Είμαι πολιτικός επιστήμων ε, για θέματα διεθνών σχέσεων και χρειάστηκα πολύ καιρό για να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό της ανθρωπιστικής δράσης υπό αυτή τη σκοπιά. Η ανθρωπιστική δράση είναι δράση αρχής. Και αυτή είναι η αρχή που αναπτύσσουμε, την αρχή της ανθρωπιστικής δράσης. Χαίρομαι που είστε εισηγητής κύριε Κεραίρο, γιατί είστε, είστε πραγματικά επαϊόν, εξηγήσετε πολύ καλά τα πράγματα και η ανθρωπιστική δράση χορηγείται όταν υπάρχει ανάγκη αρρωγής και προστασίας, είτε σε περίπτωση που οι κυβερνήσεις ε, είτε δεν είναι ικανές είτε δεν είναι πρόθυμες να παράσχουν αυτές τις, ε, ε, αυτή τη βοήθεια. Αυτή είναι η διαφορά από την ανάπτυξη από την αναπτυξιακή βοήθεια που την παρέχουμε από κοινού με τις κυβερνήσεις, συνεργασία. Οι δύο βασικές αρχές ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η αλληλεγγύη και η αμεροληψία. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες, αλλά και η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία είναι σημαντικές ε, αρχές, όπως και η πρόσβαση. Σε μια εμπόλεμη κατάσταση χρειαζόμαστε την αρχή της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανθρωπιστικής δράσης θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του πληθυσμού άσχετα από πολιτικά κριτήρια. Συμφωνώ ότι σε ένα άλλο πλαίσιο, σε μια μακροχρόνια κρίση για παράδειγμα, σε περίπτωση θεομηνίας φυσικής καταστροφής, εκεί η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και εξωτερικής δράσης. Αλλά η εξωτερική πολιτική είναι ο τρόπος που παρουσιαζόμαστε στη διεθνέ προσκήνια με βάση τις αρχές, τις αξίες μας και τους στόχους μας. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε λοιπόν την ανθρωπιστική δράση με την εξωτερική δράση. Αν πραγματικά θέλουμε να ε, χορηγήσουμε ανθρωπιστική δράση οικουμενική. Οπότε πρότεινε ξεχωριστό Συμβούλιο Υπουργών για την ανθρωπιστική δράση γιατί Ε, το θεωρώ σημαντικό παρόλο που δεν είμαι σίγουρη είναι καλό αυτό το μήνυμα που δίνουμε. Γιατί ίσως ε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ε, ανθρωπιστική δράση που στη, στη, τελική ανάλυση είναι απάντηση στις αποτυχίες και τα λάθη μας. Γιατί αν τα πράγματα είχαν γίνει σωστά δεν θα χρειαζόμασταν καν ανθρωπιστική δράση. Οπότε με ένα ξεχωριστό τέτοιο συμβούλιο ανθρωπιστικής δράσης ίσως το μήνυμα είναι λάθος. Γιατί πάντα πρέπει να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτές τις λεπτές αποχρώσεις που σας περιγράφω. Υπάρχει τάση σε μερικές διακηρύξεις, ε, πρόσφατα και του, της προσώπου προσώπου ε, για καταστάσεις όπως αυτή της Συρίας, να μπερδεύουμε την εξωτερική δράση με την ανάγκη ανθρωπιστικής δράσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να παρεμποδίσει τη, το τη δράση του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων και να αποβεί βάρος της προστασίας τους. Ερίκε. Α, συγγνώμη. Η διάσκεψη κορυφής είναι μια διάσκεψη με πολλούς φορείς, πολλούς ενδιαφερόμενους, όχι μόνο κυβερνήσεις. Βέβαια, μερικοί είπαν ότι δεν θα αναλάβουν δεσμεύσει αν δεν είναι διακυβερνητικοί. Ναι, το θέμα είναι ότι έθεσε και το οικονομικό. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Μα αυτό είναι ο λόγο. Επειδή ακριβώ δεν θα είναι οι κυβερνήσει αυτέ που θα κάνουν τι διαπραγματεύσει για τι συμφωνίε, για τι συμβιβαστικέ προτάσει, Γι' αυτό και καλό θα ήταν έχουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Σαφή συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα περιχαρακώνουν την διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έτσι εμπλέκονται άμεσα οι κυβερνήσεις. Και πότε περιμένουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Οκτώβριο, μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε την έκθεση του και τον Οκτώβριο και θα επανέλθουμε στη συζήτηση όσο πλησιάζει η ώρα και για την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη μελέτη, γιατί πραγματικά μας φωτίσατε για πολλά θέματα. Ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε στο σημείο 13, το προηγούμενο. Έχουμε σκληρή δουλειά για το απόγευμα. Έχουμε πολλά και μείζωνα θέματα. Σημείο 13, το θέμα των φύλων και της ανάπτυξης. Δεν ξέρω που είναι οι καλεσμένοι μας θα έρθουν στο Προεδρείο. Παρακαλώ οι καλεσμένοι να έρθουν να καθίσουν εδώ στο Προεδρείο ένα λεπτό για να λάβουν θέσεις. Ωραία, έχουν λάβει θέση καλεσμένοι μας. Ο λόγος που έχουμε σήμερα τη συζήτηση είναι γιατί έχουμε και στο παρελθόν συζητήσει το θέμα της, του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το νέο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη για την επόμενη πενταετία. Το θέμα των φύλων για μένα είναι πολύ σημαντικό. Οπότε δεν θέλουμε κανένα να μείνει πίσω. Σίγουρα δεν μπορούμε να αφήνουμε το μισό παγκόσμιο πληθυσμό πίσω. Γιατί με τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους και με τα μελλοντικά σχέδια δράση για την ανάπτυξη πρέπει να λάβουμε υπόψη την ισότητα των φύλων. Γιατί είναι άνηση η πρόοδος μεταξύ τους μερικές φορές. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν καλωσορίζω σήμερα τέσσερις εμπειρογνώμονες που θα μας παρουσιάσουν ε, τις ε, απόψεις τους. Πρώτα η Ντάκμαρ Σούμαχερ από την ομάδα γυναίκες των Ηνωμένων Αθηνών θα μας μιλήσει για το γενικό πλαίσιο και τις προετοιμασίες ε, εν ώψη της διάσκεψης Αντίσα Μπέμπα για την ε, χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και για τους του βιώσιμου αναπτυξιακού στόχου και τη σχετική διάσκεψη τη Νέα Υόρκη. Η κυρία Πετρούζη θα μα παρουσιάσει την αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το προηγούμενο σχέδιο δράση. Ήδη έχουμε την αξιολόγηση για το σχέδιο δράση και έχουμε και τον Ζων Λουι Βίλ. Δεν έχει έρθει ακόμη. Που θα μα μιλήσει για το επόμενο πρόγραμμα. Τα διδάγματα που αντιλήσαμε από το προηγούμενο πρόγραμμα και τι προοπτικέ του επόμενου. Και η Σεσίλ Βερνό από την Concord. από το Γερμανικό Ίδρυμα για τον Παγκόσμιο Πληθυσμό και θα μας παρουσιάσει τη σκοπιά των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τι πρέπει να περιμένουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε από το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων. Φυσικά Μα ενδιαφέρει και το χρονοδιάγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο δράση. Αλλά ήταν, ήταν πολύ σύντομο αυτό το χρονοδιάγραμμα. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα υποβάλει το, την πρόταση για το σχέδιο δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ζητήσει από το Συμβούλιο ήδη τον Οκτώβριο να καταλήξει συμπεράσματα. Πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είναι απαράδεκτο ένα σχέδιο δράση να προ, προβάλλεται ω έγγραφο εργασία απλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπρεπε να γίνουν διαβουλεύσει, να γίνει μια πιο εκτενή διαδικασία. Αλλά ίσω είναι αυτή προοπτική και αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον θα έχουμε ευκαιρία για συζήτηση και ψήφισμα στην Ολομέλεια. Όχι έκθεση πρωτοβουλία, γιατί πρώτα πρέπει να δούμε γραπτός, τη γραπτή πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά δεν θα έχει μείνει χρόνο. Πάντω είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα για μα. Θα ανταποκριθούμε στι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να μην χρονοτριβάλλω, θα δώσω το λόγο στην κυρία Σούμαχερ για να μα πει τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά θα περάσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Dagmar αν μπορεί να τηρήσει και το πεντάλεπτο, θα σου ήμουν ευγνώμων. Um, Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ για την παρουσία μου εδώ. Είναι εξαιρετική η κατάσταση για να το συζητήσουμε παγκόσμια, αλλά και το τι γίνεται στην Ευρώπη με το πρόγραμμα δράση για την ισότητα των φύλων. Έχουμε όμως και κάποιες ε, δραστηριότητες που μας ε, ενθαρρύνουν. Για παράδειγμα έχουμε την συνάντηση κορυφή στην Αντισαμπέμπα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να επιτύχει αυτή η συνδιάσκεψη. Ε, χαιρόμαστε για τα κείμενα που έχουμε ήδη δει για την ισότητα των φύλων και το σωστό λεξιλόγιο. Επίσης έχουμε και ένα πλαίσιο. Χαιρόμαστε για τους αυτόνομους στόχους και τη στήριξη της Ένωσης γι' αυτό. Και επίσης το mainstreaming στους άλλους στόχους, δηλαδή στην περίπτωση πάντα των θεμάτων ισότητας των φύλων. Θέλουμε συγκεκριμένους στόχους με δείκτες για την ισότητα των φύλων σε όλους τους άλλους στόχους. Και όλοι οι συνάδελφοι εργάζονται πολύ σκληρά γι' αυτό. Και επίσης Έχουμε και το ΚΑΠ 21 κόπ 21 τη συναντηση COP21 βεβαίως. Πρέπει να επιτύχει. Γιατί αν δεν επιτύχει, δεν θα επιτύχει το θεματολόγιο της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Και έχουμε και την αναθεώρηση του ρόλου των γυναικών στην ασφάλεια και την ειρήνη ε, μετά από 15 χρόνια που θα υποβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και τα κράτη-μέλη και συνολικά και εσείς έχετε συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία και θέλουμε ισχυρές δεσμεύσεις από τα κράτη-μέλη. Ούτως ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε επιτύχει αρκετά, τουλάχιστον να έχουμε κάνει μια αποτίμηση του που βρισκόμαστε. Έχουν σημειωθεί μεγάλες πρόοδοι στην ε, νομοθεσία, αλλά πραγματικά να αλλάξει η ζωή των γυναικών, να προσεγγίσουμε την ε, ισότητα των φύλων, δεν έχουμε κάνει τόσο πολλά. Όπως λέει ο Γενικός μου Διευθυντής, σε καμία χώρα δεν υπάρχει απόλυτη ισότητα των φύλων. Επίσης, στις 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τη συνάντηση κορυφής για δεσμευτικές υποσχέσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ, όπου θα πρέπει να μας πούν πώς θα εφαρμόσουν αυτά που δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί από το πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν σταθερές δεσμεύσεις για να καλυφθούν τα κενά. Κάνουμε λοιπόν έκκληση και προς την Ένωση και προς τα κράτη-μέλη να κάνουν θαραλές, να αναλάβουν θαραλές και ισχυρές δεσμεύσεις. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά αναγενιά για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων. Ξέρετε, θα έχετε ακούσει ότι έχουμε ακόμη ορισμένα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις και για την ε, διάσκεψη της Αντίσα Μπέμπα και για άλλα θέματα δεν έχουν προχωρήσει. Η Αμίνα Μοχάμεντ ήταν χθε εδώ και έκανε έκκληση για να δεσμευθεί αποφασιστικά η Ένωση για το 0,7 αναπτυξιακή βοήθειας. Και ελπίζω το Κοινοβούλιο να βοηθήσει πολύ σε αυτό. Να είναι πραγματικά ο κρούο τον κόδωνα του κινδύνου εάν υπάρξει πρόβλημα και για την επίτευξη του στόχου και μετά για την εφαρμογή του. Τώρα για την λογοδοσία και τα μέσα εφαρμογής. Νομίζω ότι θα παίξουμε ε, μεγάλο ρόλο για την επίτευξη του στόχου 5 των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων και για την ετήσια ε, επανεξέταση για το πόσο προχωρεί η επίτευξη αυτού του στόχου. Και εδώ λοιπόν θα χρειαστούμε ιδιαίτερα την στήριξη του Κοινοβουλίου. Τώρα να σας μιλήσω λίγο για τη σωστή συμπερίληψη στους προπολογισμούς των θεμάτων ισότητας. Μίλησα για την ε, συνδιάσκεψη της Αντισαμπέμπα. Θέλουμε να υπάρξει ισχυρή δέσμευση ότι θα υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση γιατί η αναθεώρηση του Πεκίνου συνήκωση απέδειξε ότι μέχρι στιγμής οι πόροι που δαπανώνται για αυτούς τους στόχους δεν επαρκούν για την επίτευξη του προγράμματος δράσης του Πεκίνου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ανανέωση της δέσμευσης των χωρών για την επίτευξη αυτού του στόχου. Έχουμε συνεργαστεί με 73 χώρε, με τα αντίστοιχα υπουργεία, για να προωθήσουμε αυτό το στόχο. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαμε την τελική συζήτηση πριν από δύο εβδομάδε εδώ στι Βρυξέλλε γι' αυτό. Συνεργαζόμεθα με του υπουργού οικονομικών, ούτω ώστε οι προπολογισμοί να λαμβάνουν υπόψη τα θέματα φύλου. Και αυτό πρέπει να υπάρξει και του επόμενου μήνε στα διάφορα παγκόσμια πλαίσια που το συζητάμε. Και αυτό που έχει υπόψη η Επίτροπο Γεωργίευα αλλά και η κυρία Τζούροβα για ε, τα κονδύλια στου προπολογισμού. Και ένα θέμα ακόμη για το πρόγραμμα δράση για την ισότητα των φύλων. Νομίζω είναι ιστορική ευκαιρία τώρα. Λόγω του ότι έχουμε αυτό το νέο διεθνέ πλαίσιο, που θα είναι σε ισχύ πριν το τέλος του χρόνου για να έχουμε ένα αποφασιστικό πρόγραμμα δράσης για την ισότητα των φύλων και για να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση στα πλαίσια των πόρων που διατίθεται για την αναπτυξική βοήθεια. Να προωθήσουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα για την ισότητα και επειδή είναι ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τους αναπτυξιακούς ε, βιώσιμους στόχους η στρατηγική για την ισότητα των φύλων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχου. Να λαμβάνονται υπόψη δηλαδή περισσότερο τα θέματα ισότητα των φύλων εντό τη Ευρώπη, αλλά και εκτό. Νομίζω ότι υπόθηκε και χθε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία το ότι το πλαίσιο αυτό θα είναι παγκόσμιο για την Ευρώπη, ιδιαίτερα για θέματα ισότητας φύλων, γιατί θέματα για παράδειγμα όπω η βία κατά των γυναικών η εργασία φροντίδας, η μη αμοιβόμενη, αντιμετώπιση των στερεοτύπων φύλων. Είναι θέματα και στην Ευρώπη αυτά και σαν αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι λοιπόν παγκόσμια αυτή η στόχη σε όλο τον πλανήτη πρέπει να εφαρμοστούν, να επιτευχθούν. Ευχαριστώ Ντάγμαρ, λέει η Πρόεδρος, για το πόσο συγκεκριμένοι ήσουν και γιατί μας είπε τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Να δώσω τώρα το λόγο στη Φεντερίκα Πετρούτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα κάνει μια ανασκόπηση της αποτίμησης του τελευταίου προγράμματος ε, δράσης ε, για την ισότητα των φίλων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η αξιολόγηση στην μονάδα ΤΕΦΚΟ της ε, Διεύθυνσης για την αξιολόγηση της ε, ισότητας των φύλων καθώς και της χειραφέτησης των γυναικών σε χώρες εταίρους για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007 με 2013. Οπότε θα σας δώσω μια σύντομη εικόνα των ε, κυρίων πορισμάτων και των συστάσεων που προέκυψαν από αυτήν την αξιολόγηση. Εν γέννη, η αξιολόγηση καταλήγει ότι ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα επιτέχθησαν, αλλά ήταν τμηματικά και δεν ήταν καλά τεκμηριωμένα. Με κάποιες λίγες εξαιρέσεις, οι αντιπροσωπείς δεν υιοθετούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να συνδυάζει το mainstreaming των φίλων και τον πολιτικό διάλογο που ήταν στην βάση του προηγούμενου GAP. Βασικό μας πόρισμα λοιπόν είναι αυτό που κινείται γύρω από τα 5 C. Ε, δεσμεύση, αφοσίωση, ε, κατανόηση του, ε, του πλαισίου, συντονισμός, χρήματα, για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε λοιπόν την απόδοση της, εξωτερι... της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης όσον αφορά τη δέσμευσή μας και την αφοσίωσή μας στο θέμα της ισότητας των φύλων. Αυτό δεν έγινε στην πραγματικότητα. Υπήρχε έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στο κεντρικά γραφεία και τις αντιπροσωπείες και γι' αυτό οι συνάδελφοι δεν είχαν κατανοήσει πλήρως ε, το περιεχόμενο της πολιτικής στήριξης της ισότητας των φύλων και τη σημασία του για την αναπτυξιακή συνεργασία. Σε σχέση με τις δυνατότητές μας τις ικανότητές μας η οικονομική δέσμευση για την πρόθεση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στην περίοδο αυτή ήταν αυξημένη. Όμως Ε, δεν ακολουθήθηκε το ίδιο μονοπάτι όσον αφορά το, το δυναμικό. Η διοίκηση θεώρησε πως ε, το προσωπικό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει βασικά το, να αντιμετωπίσει το θέμα μόνο με το άτομο το οποίο έχει αναλάβει το θέμα του φίλου στις αντιπροσωπείες. Ε, ε, το συγκεκριμένο άτομο συνήθως είναι νεαρό, είναι αρχάριος υπάλληλο, οπότε δεν έχει συνήθως τις δυνατότητες πραγματικά να δράσει. Άρα λοιπόν ε, τελικά το θέμα του φίλου δεν θεωρήθηκε ως κοινή ευθύνη. Και τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν αφήνονται περισσότερο σε ατομική προσήλωση και όχι σε οργανωτικό αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά τα χρήματα ε, cash για την ισότητα των φύλων, η οικονομική συμβολή και η δέσμευση για την περίοδο αυτή έχει αυξηθεί από 1,6 εκατομμύρια το 2007 σε 311 εκατομμύρια το 2011. Ωστόσο, Κατέστη δυνατόν να καθοριστεί λοιπόν η δημοσιονομική συμβολή ε, μόνο για δράσεις ε, συγκεκριμένα υπέρ της ισότητας των φύλων. Όμως για το mainstreaming οι εμπειρογνώμονες δεν μπορούσαν να έχουν συγκεκριμένα ποσά λόγω στην ισχνή εφαρμογή του σηματοδότη για το φύλλο που είναι αυτό το εργαλείο, το μέσο το οποίο έχει αποφασιστεί μέσω του ε, του οδηγού του όσα. Υπάρχουν όμως ε, σημαντικές ε, χρήσεις της ανάλυσης των φύλων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε προγραμματισμό και οι δείκτες αυτοί ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται καταλήλως μέσα στο γενικότερο πλαίσιο δικτών για την αξιολόγηση του κάθε προγράμματος. Πάντως το φύλλο δεν είναι σαφώς ε, ενσωματωμένο στη στρατηγική αναχώρα ούτε σαφώς περιέχεται στους δείκτες. Ως αποτέλεσμα λείπει από τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων και σε στρατηγικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά το GAP. Τα αποτελέσματα δεν είναι επαρκή σε σχέση με τα νούμερα που έχουμε στα χέρια μας και δεν υπάρχει καμία προβλεπόμενη κύρωση εάν κάποια αντιπροσωπεία δεν δώσει έκθεση για τα θέματα ισότητας των φύλων. Και αυτό βεβαίως ήταν ένα πρόβλημα όσον αφορά την λογοδοσία και οι εκθέσεις για το φύλλο δεν ενσωματώνονται στην έκθεση εξωτερικής δράσης ε, του γραφείου, που είναι το βασικό, η βασική αναφορά που συντάσσουν οι αντιπροσωπείες προς ε, τα κεντρικά Τώρα, για το συντονισμό δεν υπάρχει μεγάλη κατανόηση όσον αφορά το πλαίσιο και τη χρήση της πολιτικής ανάλυσης ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα προγράμματα αλλά και τον διάλογο ως αποτέλεσμα με κάποιες μικρές εξαιρέσεις βεβαίως γιατί υπήρξαν και καλές ε, πρακτικές από κάποιες αντιπροσωπείες όπως ε, το Μαρόκο, η Αιθιοπία και το Αφγανιστάν με λίγες λοιπόν εξαιρέσεις οι αντιπροσωπείες δεν έχουν σαφή εικόνα ε, όσον αφορά τις ευκαιρίες που υπάρχουν για την ισότητα των φύλων, για να ενημερώσουν δηλαδή την στρατηγική αναχώρα, αλλά ούτε και την αντίστοιχη επιτροπή, καθώς και τη στρατηγική συνεργασία με την, ε, ε, ε, με την κυβέρνηση εταίρο, με τις μικιό, τους διεθνείς οργανισμούς και τους διεθνείς εταίρους. Αυτά είναι τα συμπεράσματα. Τώρα όσον αφορά τις συστάσεις, θα σας τις παρουσιάσω σύντομα. Η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να ηγηθούν όσον αφορά την ανάπτυξη μια συνέχιση θα δοθεί στον ΚΑΠ, όπω αυτό έχει ζητηθεί από το Συμβούλιο. Και αυτό σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη, γιατί αυτή είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλλον αυτό ο συντονισμό είναι πολύ μεγάλη σημασία. Αργότερα θα ακούσετε και μια εικόνα για το τι κάνουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη σύσταση. Η Κομισιόν και η εξωτερική δράση, διότι οι συστάσεις πάντοτε απευθύνονται προς την Κομισιόν και προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα πρέπει να βρουν ρυθμίσεις ε, για να μπορέσουν να επιτύχουν την ισότητα των φύλων αλλά και να μπορέσουν να αποδώσουν σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης καθώς και την συμπληρωματικότητα με τα κάτι μέλ. Πάντοτε προς την Κομισιόν και την εξωτερική δράση θα πρέπει να φτιάξουν μια ξεκάθαρη ρύθμιση για να μπορέσουν να επιτύχουν την ισότητα των φύλων Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκλήρηση ε, της έκθεσης ε, λογοδοσίας προς ε, τα βασικά μέσα αναφοράς όπως τα ανέφερα και προηγουμένως. καθώς και επίσης με το σύστημα παρακολούθησης και, την, και και την ομάδα για την βελτίωση της ποιότητας, θα πρέπει όλα αυτά να συνδυαστούν μεταξύ τους και να ενισχυθούν. Οι αντιπροσωπείες αλλά και οι πρεσβείες των κατορμελών θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα και να επενδύσουν στην ανάλυση της ε, ισότητας των φύλων γιατί αυτή η ανάλυση βρίσκεται στη βάση της στρατηγικής και χωρίς σωστή ανάλυση δεν μπορούμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένους δείκτες που είναι βεβαίως οι πιο σημαντικοί ώστε να υπάρχει η λογοδοσία, να υπάρχει η παρακολούθηση και να μπορέσουμε τελικά να έχουμε αποτελέσματα στο τέλος. Ε, η πρόεδρος διακόπτη. Ε, καλύτερα να κλείσετε γιατί ο χρόνος σας τελείωσε, διακόπτη πρόεδρος. Νομίζω ότι τα βασικότερα μηνύματα ήδη τα ανέφερα. Συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Τρία λεπτά είχατε στη διάθεσή σας. Πάντως, όπως είπε και ο Ενρίκε Γκερέρο, συνήθως οι βουλευτές έχουν δύο λεπτά στην Ολομέλεια. Οπότε έχουν συνηθίσει να περνάνε το μήνυμα σε λίγα λεπτά ήρθε και ο Ζόλι Βίλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπα ότι θα πρέπει να μας ε, πείτε το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη νομική ισχύ, τη νομική φύση των εγγράφων, γιατί από ό,τι κατάλαβα πρόκειται για έγγραφο εργασία με συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Θέλουμε λίγο χρόνο για να δούμε ποιο θα είναι το πόνιμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης. Ε, πολύ σύντομο χρονοδιάγραμμα μας υποβάλλατε. Πάντως ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ήταν πολύ ειλικρινής ε, στην αποτίμηση του προηγούμενου προγράμματος. Τώρα έχουμε το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων. Και ε, πήγαμε στην αντιπροσωπεία και στο αρμόδιο γραφείο μας είπαν ότι δεν υπάρχει αρκετή επικοινωνία. Και μάλιστα ε, είχαμε, θα έχουμε το Σεπτέμβριο τους ε, επικεφαλής αντιπροσωπείων όλων των γραφείων, αλλά δεν ε, είναι όλοι ενήμεροι για θέματα ισότητας φύλων. Θα πρέπει αυτό το θέμα να συνεκτιμάται παντού. Ακούσαμε το πρόβλημα με την λυπή δεδομένα που δίνουν οι αντιπροσωπείες. Τι θα αλλάξει, ποιο θα είναι το καινούργιο στοιχείο του νέου σχεδίου δράσης, ποια θα είναι η διαδικασία, παρακαλώ. Ευχαριστώ και συγγνώμη που Χρειάστηκε να έρθω τρέχοντας. Τελευταία στιγμή ήρθα πάντως, αυτό είναι σημαντικό. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός και να απαντήσω σε ερωτήσεις. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και ε, την πρόσκληση προς εμένα αλλά και προς τους συναδέλφους γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ευρύ ανάλυση και σωστό απολογισμό. Αναφέρθηκε ότι το GAP 2010-2015 περιλαμβάνει εξολόγηση και δύο κρατών μέλων δεν ήταν μόνο αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και αξιολόγηση Ισπανίας και κάτω χωρών. Οπότε ήταν σημαντικό να γίνει μια κοινή προσπάθεια και ευχαριστώ θερμά και τις δύο χώρες που ανέλαβαν αυτές τις προκλήσεις και ανταπεξήλθαν. Για τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αλφαβήτα τρόπο βρίσκεται κοντά στην υιοθέτηση του επόμενου σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων και ε, το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης κατέληξε συμπεράσματα ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ένα εύρωστο νέο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2016-2020. Οπότε τώρα από πολιτική άποψη θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει τι μορφή θα δώσει σε αυτό το σχέδιο δράσης. Τη μορφή της ανακοίνωσης ή του εγγράφου εργασία. Δεν έχουμε οριστικοποιήσει ακόμη, δεν έχουμε αποκρισταλώσει τη γνώμη μα. Δεν αποκλείται να είναι και έγγραφο εργασία, αλλά δεν είναι σίγουρο. Όποια απόφαση πάντω και ληφθεί, η διαδικασία θα, πρέ... θα προβλέπει η υιοθέτηση γύρω από τον Ιούλιο, ανάλογα με το πότε που θα ξεκινήσει, γύρω στα μέσα Ιουλίου, 10-20. Οπότε το χρονοδιάγραμμα είναι σχετικά σαφές. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία έχει δείξει προθυμία και ζέση ώστε να συζητηθούν τα έγγραφα και να υιοθετηθούν τα συμπεράσματα στο επόμενο Συμβούλιο Ανάπτυξης που θα λάβει χώρα στα τέλη Οκτωβρίου. Οπότε αυτό θα είναι και το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες. Και μάλιστα την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ίσως ε, υιοθετηθεί και από εμάς, ίσως και λίγο νωρίτερα, ίσως λίγο αργότερα. Πάντως, αν γίνει έγκριση τον Ιούλιο ή αρχές Σεπτεμβρίου, θα απομείνουν δύο μήνες από την έγκριση μέχρι τα προβλεπόμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Όλα αυτά βρίσκονται υπό συζήτηση ακόμη, γιατί τώρα αρχίζει τις προεργασίες η Λουξεμβουργιανή Προεδρία για το δικό της εξάμενο. Πάντως, αν δεν εγκριθεί εν αυτό το χρόνο το χρονοδιάγραμμα, το σχέδιο δράσης, δεν θα προλάβει και το Συμβούλιο να εκδώσει τα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο. Επί τη ουσία. η Φεντερίκα έκανε μια πολύ καλή ανακεφαλαίωση των βασικών συμπερασμάτων της αξιολόγησης και ευχαριστώ θερμά τους αξιολογητές για την έκθεση που εκπώνησαν. Δυστυχώς ε, είχαμε πολλά κενά σε ό,τι αφορά την ε, δέσμευση και την προσήλωση σε διάφορα επίπεδα. Γιατί δυστυχώς είναι ουραγή τα ζητήματα του φίλου για, πολλούς, ε, για πολλές αντιπροσωπείες και πολλοί επικεφαλείς αντιπροσωπιών αδιαφορούν για το θέμα των φύλων, της ισότητας των φύλων και δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ανάγκη συνεκτίμηση τη διάσταση φύλου σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα. Πολλές φορές το υπενθυμίζουμε, αλλά δεν εισακούγεται πάντα το έτοιμά μας. Πάντως από την αξιολόγηση η Φεντερίκα ε, στάθηκε στο θέμα της έλλειψης ανάλυσης. Μερικές χώρες δεν έχουν καν αυτή την ανάλυση υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων. Οπότε για συγκεκριμένα προγράμματα δεν έχουμε ιδέα για το πώς έχει η κατάσταση της ισότητας των φύλων και στο μελλοντικό σχέδιο δράσης αυτό θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή να έχουμε υποχρεωτική ανάλυση υπό το πρίσμα του φύλου στα προγράμματα αυτά για να διαμορφώσουμε μία εικόνα. Γιατί πώς αλλιώς θα καταμετρήσουμε την πρόοδό μας. Επίσης, θέλουμε σωστή εφαρμογή και διεξοδική των δικτών του φύλου για την ισότητα των φύλων. Γιατί οι στόχοι ήταν ε, πολύ πιο φιλόδοξοι και προσδοκίες από τα αποτελέσματα. Είχαμε στόχο το 75% προγραμμάτων που θα λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των φύλων και στο τέλος περίοδου μόνο το 39% καταφέραμε. Βέβαια καλύτερο από το 18% που είχαμε στην αρχή, αλλά παρόλα αυτά πόρο απέχουμε από τον αρχικό μας στόχο που ήταν το 75%. Αλλαγή της εντολής των επικεφαλής αντιπροσωπιών που είχαν λάβει την οδηγία να συμπεριλάβουν το θέμα της ισότητας των φύλων στα προγράμματα. Επίσης, ομάδα στήριξης ποιότητας στην αξιολόγηση και προετοιμασία της απόφασης. Να γίνεται συστηματική προώθηση και αναφορά για το θέμα της ισότητας των φύλων στα διάφορα προγράμματα και να βελτιώσουμε το σύστημα παρακολούθησης των σχεδίων μα με συνεκτίμηση τη διάσταση του φύλου. Θα πρέπει να εκπαιδεύουμε του αξιολογικέ και του αξιολογητές και τους ελεγκτές ε, και να του ευαισθητοποιήσουμε στο θέμα τη ισότητα των φύλων και τη συνεκτίμηση τη. Θέλουμε πραγματικά ε, θεσμικέ αλλαγέ που θα πρέπει να προηγηθούν. Τώρα, επί τη ουσία, το νέο σχέδιο δράση για την ισότητα των φύλων θα υιοθετήσει μια τρίπτυχη προσέγγιση, σωματική βία, η σωματική ακαιρεότητα, βία πάσης φύσεως, η οικονομική χειραφέτηση, δεύτερος πυλώνας, δεύτερος άξονας και τρίτον οι φωνές που λέμε, ε, εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ε, πολιτικό, οικονομικό και ούτω καθεξής. Φυσικά δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για όλους. Θα πρέπει κάθε αντιπροσωπεία να κάνει την ανάλυση, να αξιολογήσει την κατάσταση στη δεδομένη χώρα και να δει το gap το σχέδιο δράση υπό το πρίσμα των διαφόρων στόχων και να εξετάσουμε τον αντίκτυπό τους και τι μέτρα θα λυθούν. Το θέμα είναι πώς θα γίνει η καταμέτρηση της πρόοδου και πώς θα δώσουμε μια συνέχεια στις δράσεις ή πώς θα κάνουμε την ενημέρωση για τις δράσεις. Πάντως έχουμε πολλές καλές προτάσεις σχετικά η Γκάνα και το Μαλάουι φυσικά δεν θα υιοθετήσουν τις ίδιες λύσεις, γιατί κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Αλλά αυτό θα το κρίνουν οι αντιπροσωπείες. Αυτά και βάζω τελεία, γιατί βλέπω ότι έχω παραβίδει το χρόνο μου. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα πρέπει όχι μόνο να έχουμε αποφάσεις ε, του Συμβουλίου, αλλά να υπάρχει και κοινοβουλευτικός έλεγχο Διότι αυτή είναι η συνήθις διαδικασία, δηλαδή όταν το, η Επιτροπή εγκρίνει μια πρόταση περνάει και από το Κοινοβούλιο για να υπάρξει έλεγχος και είναι εξάμεινο. Δεν θέλουμε λοιπόν μόνο αποφάσεις του Συμβουλίου αλλά και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Λοιπόν η Σασίλ θα μας πει τώρα για το πρόγραμμα Concord. Ευχαριστώ. Έχουμε ενώπιον μας την DISABEBA και το νέο πρόγραμμα δράση και τη Νέα Υόρκη από πλευρά τη ομάδα εργασία Concord για την ισότητα των φύλων θα είμαι πολύ σύντομη. Αλλά μετά στη συζήτηση μπορούμε να δούμε περισσότερα τα θέματα. Όλα όσα λέω ισχύουν και για την Άντις και για την Αντισαμπέμπα. Ε, Έχουμε λοιπόν ε, τριπλή προσέγγιση, mainstreaming του φύλου, στοχευμένες δραστηριότητες και πολιτικό διάλογος. Αλλά δεν υπάρχει δέσμευση για την εφαρμογή του προγράμματος. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αξιοποιήσει ως ευκαιρία για να παίξει ηγετικό ρόλο, να μην είναι μόνο ένα κείμενο των υπηρεσιών, να είναι η Ένωση. Και χρειάζεται και διαθεσμικός διάλογος, διοργανικός με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Λοιπόν, το πρώτο, όπως είπα, είναι να διευρυνθεί η προσέγγιση μας όχι μόνο για την ανάπτυξη, συνολικότερα για την εξωτερική δράση, είτε είναι ανθρωπιστική βοήθεια, ειρήνη, ασφάλεια κτλ. Αυτό σημαίνει να συνεργαζόμεθα περισσότερο με τα κράτη-μέλη και πρέπει να δούμε και τα ίδια τα προγράμματα. Με κριτικό μάτι υποστηρίζουμε αυτά που έχουν ε, στο κέντρο των προσπαθειών τους ε, την ισότητα των γυναικών. Πρέπει να προσαρμοστούμε λοιπόν. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση εξάντε όταν για παράδειγμα έχουμε εταιρικές σχέσεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει προσέγγιση και ε, ο τρόπος λειτουργίας των θεσμικών οργάνων πρέπει να δεσμευθούν όλοι. Μερικές ιδέες της Κομισιόν δείχνουν ότι το έχουν σκεφτεί το θέμα και το στηρίζουμε. Να είναι στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας και όχι απλώς να λέμε «α, το κάναμε γι' αυτό και να βάλουμε ένα χι δίπλα». Πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση και πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται πόροι. Χρειάζονται πόροι. Πρώτα απ' όλα προσωπικό. Αλλά και περισσότερες δυνατότητες. Ε, καλύτεροι, καλύτεροι εργαζόμενοι. Δηλαδή και καλύτερη οργάνωση και να έχουν δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους δείκτες για ισότητα των φύλων. Άρα δεν είναι μόνο θέμα να δούμε πόσες γυναίκες σε ποια θέση, αλλά να δούμε ανατομή. Για παράδειγμα για την ενέργεια, ας πούμε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για την ενέργεια. Τι θα προωθήσει σε αυτή τη χώρα, σε ποιο πλαίσιο, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Πρέπει να δούμε και πέρα από τις γενικές στατιστικές. Και να δούμε και ποιες ομάδες ακριβώς. Οι ομάδες, ε, οι γυναίκες δεν είναι όλες μια ομάδα. Ορισμένες, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν άλλα στοιχεία που τους κάνουν πιο ευάλωτες. Μπορεί να είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρέπει να δούμε όλες τις ε, ε πλευρές και σεξουαλικό προσανατολισμό. Και φυσικά μετά είναι και η οικονομική πόροι. Θέλουμε η Ένωση να δεσμευθεί και στην Αντισαμπέμπα για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αν δούμε μέχρι πού θα πάει μέχρι το 2050 η αναπτυξιακή μας βοήθεια, δεν λέγονται πολλά για στοχευμένη δράση. Μόνο 1,5 ή 1,75 θα αφορά τις δράσεις για την ισότητα των φύλων. Άμα δούμε και την διμερή συνεργασία, σε καμία χώρα που έχει διμερή συνεργασία με μια άλλη δεν, είναι, δεν υπάρχει εστίαση στην ισότητα των φύλων. Κάπου λέγεται ότι το φύλλο, η ισότητα των φύλων πρέπει να είναι προτεραιότητα, αλλά πώ θα γίνει αυτό, χρειάζονται καθεντήρε γραμμέ και χρειάζεται και λογοδοσία γι' αυτό. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη γι' αυτό. Άρα έχει να κάνει με το πόσο αυτοί οι οποίοι είναι στα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της χώρας έχουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη. Και τέλο, για την χρηματοδότηση εκπαίδευση. Η αναπτυξιακή βοήθεια είναι μόνο ένα τμήμα, αλλά έχει καταλητικό αποτέλεσμα. Θα θέλουμε να το δούμε. Θέλουμε να ενισχύσουμε μερικά βασικά στοιχεία. Η προσέγγιση μας πρέπει να βασίζεται στα δικαιώματα. Έτσι θα βοηθήσει και η αναπτυξιακή βοήθεια. Συμφωνώ λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πόσοι συμμετέχουν στα διάφορα όργανα αλλά και στην οικονομία. Και να είναι ε, αυτό ορατό στα στοιχεία που συλλέγουμε. Να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στη σεξουαλική υγεία και την πρόληψη και να επιτύχουμε αυτή την ισότητα μεταξύ των φίλων. Και θέλουμε ισότητα των φίλων με την ευρύτερη έννοια. Να συμπεριλαμβάνονται όλε τι σεξουαλικές μειονότητε, για παράδειγμα. Ο δεύτερος ρόλος της Ένωσης είναι να παίξει ρόλο στον πολιτικό διάλογο με τις χώρες με τις οποίες έχουμε εταιρική σχέση και να υπάρχει ε, ευθυγράμμιση και με τους στόχους για ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τα βασικά αίτια της ανισότητας των φύλων. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να επηρεάσουμε σε κάθε τομέα. Και συμφωνώ με αυτό που πει οι χώρες εταίροι πρέπει να συμπεριλάβουν στους προπολογισμούς τους τα κονδύλια για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε ε, να σχεδιάσουν σωστές δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές. Κανένας ε, φόρος δεν είναι ουδέτερος από πλευράς φύλου. Οι γυναίκες κυρίω δουλεύουν στην άτυπη οικονομία. Και αυτές αγοράζουν τα βασικά προϊόντα για την οικογένειά του. Αν αυξήσει το ΦΠΑ για παράδειγμα θα επηρεάσει κυρίω τις γυναίκες. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε πώ γενικά ο προπολογισμό λαμβάνει υπόψη το φύλλο και να κάνουμε συγκεκριμένε ενέργειε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό και είναι μία από τις βασικές συνταγές για να αυξηθούν οι πόροι για την ισότητα των φύλων στους ε, ε, δημόσιους προπολογισμούς. Και τέλος, λογοδοσία. Λογοδοσία. Λογοδοσία. Είναι κλειδί. Μπορεί να έχουμε τα καλύτερα σχέδια, όπως είδαμε στο προηγούμενο γκάπ, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε αν εφαρμόζονται. Βεβαίως θέλουμε και οι στόχοι για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη να είναι ρεαλιστικοί Θέλουμε όλοι οι δείκτες να συνδέονται στο παγκόσμιο πλαίσιο, να έχουμε σωστά στοιχεία υψηλού επίπεδου, να δούμε και την κατανομή αναηλικία. Για παράδειγμα δεν έχουμε καθόλου στοιχεία για τις ομάδες ηλικία 10 με 14 και πάνω από 50. Και πάνω από 50 υπάρχει ζωή, ξέρετε. Και επίσης πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία. Πώς τα χρησιμοποιούμε για την παρακολούθηση της εφαρμογής. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει, για παράδειγμα, μια δημόσια παρουσίαση από τι χώρε ποιε είναι οι προτεραιότητες του για να δούμε μετά πόσο τι εφαρμόζουν αυτέ τι προτεραιότητες. Να αποφασίζουν οι χώρε για τι προτεραιότητες του με βάση τι συνθήκε τη χώρας αυτέ. Εμεί απλώ να ξέρουμε ποιε είναι για να παρακολουθούμε μετά τι εφαρμόζουν. Γι' αυτό θέλουμε να είναι δημόσια τα στοιχεία, μηχανισμού λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνέ. Και όλα αυτά χρειάζονται Πολύ στήριξη, πολύ προσωπικό, καταλήγοντας. Λοιπόν, όλες οι οργανώσεις γυναικών αυτή τη στιγμή δεν έχουν επαρκείς πόρους. Πρέπει να αυξηθεί λοιπόν η στήριξη για όλες τις οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα γυναικών για να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα δράσης. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βήματα ενώπιόν μα και προσβλέπω και στην περαιτέρω συζήτηση και ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Ακούσαμε το παγκόσμιο πλαίσιο, την αξιολόγηση του προηγούμενου σχεδίου δράση για, την ισότητα των φύλων, το επόμενο και τη γνώμη των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τώρα, η Χάιντι Χάουταλα που πρωτοστατεί στην Επιτροπή ε, και είναι αρμόδια για τα θέματα των φίλων. Θα σας σοκάρω, αλλά νομίζω ότι όσοι ασχολείται με την ε, αναπτυξιακή συνεργασία ε, και την εξωτερική δράση θα πρέπει να το τιμωρούμε με ηλεκτροσόκ όταν ξεχνάει τα θέματα του φίλου. Μπορεί να σας σοκάρω, νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε. Έχουν περάσει δεκαετίες και πολύ εύκολα ξεχνάει κανείς το θέμα της ισότητας των φίλων. Και ε, μερικές φορές ξεχνάμε τα γυαλιά μας, στο φακό με το μέσα από τον οποίο βλέπουμε και τα θέματα των φίλων. Και όταν βάζουμε αυτά τα γυαλιά βλέπουμε πόσο σεξουαλική βία υπάρχει, σεξιστική βία εις βάρος των γυναικών. Ξέρω ότι υπάρχει και σεξιστική βία εις βάρος των ανδρών. Έχω ακούσει από τρόπε ιστορίες για σεξουαλική βία που έχουν υποστεί. Είναι θέμα φίλων. Ε, γάμοι παιδιών, καταναγκαστική γάμοι, απαγόρευση, η άρνηση έκτρωση υπό ασφαλείς ε, συνθήκες και ο οικονομικός παράγοντας. Όλοι, από την Παγκόσμια Τράπεζα μέχρι τις γυναίκες των Εθνών, μπορούν να μας αποδείξουν με χιλιάδες τρόπους πόσο μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη επενδύοντας στα κορίτσια και στις γυναίκες. Γιατί λοιπόν δεν με και αυτή τη σκοπιά σε αυτό το σούπερ έτος ανάπτυξης που είναι το 2015 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, Ελπίζαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ήταν πιο φιλόδοξη. Γιατί έχουμε πολλά καλά συστατικά. Καταρχήν την αξιολόγηση. Τι προηγούμενε δεκαετίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χαρακτήριζε εμπιστευτική αυτή την αξιολόγηση γιατί είναι επέσχυντο ε, να διαπιστώνουμε τι αδυναμίες υπάρχουν σε επίπεδο δράσεων ακόμη ε, και λόγων και τα κενά που υπάρχουν. Και ελπίζω το νέο σχέδιο δράση να λάβει τη μορφή ανακοίνωση προ όλα τα θεσμικά όργανα και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί, όπω είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι κάτι που απευθύνεται μόνο στα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο. Επίση, ε, ήταν σαφέ και ακούσαμε και από προηγούμενε συζητήσει ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερα θέματα. Θέματα έχουμε αρκετά για την ισότητα των φύλων. Αλλά θα πρέπει να περιλάβουμε μηχανισμούς, ε, λογοδοσία, οικονομικούς μηχανισμούς για χρηματοδότηση. Αυτό χρειαζόμαστε. Θέματα έχουμε. Και πραγματικά, ίσως θα πρέπει να απειλούμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο ε, σε περίπτωση που αμελήσει ξεχάσει το θέμα της ισότητας των φύλων, να τους απειλήσουμε με ηλεκτροσόκ. Ελπίζω να μην είναι πολύ ε, βίαιη η πρότασή μου. Επίση, διαπιστώνω ότι μπορούμε κάλλιστα να συμπεριλάβουμε την ισότητα των φύλων στον προγραμματισμό μα και στον προπολογισμό. Και μάλιστα είχα την τιμή να λάβω μέρο πρόσφατα σε ένα σεμινάριο στι Βρυξέλλες με θέμα αύξηση τη χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων. Κοινή εκδήλωση ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών και κάποιων άλλων οργανώσεων. Και εκπρόσωποι τη Βολιβίας και άλλων αντισωμένων χωρών μα εξηγούσαν τι κάνουν ε, οι χώρες και οι Υπουργοί Οικονομικών για τα θέματα αυτά. Και όπως είπε η κυρία Βερνάου, και οι κυβερνήσεις των εταίρων μας θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτό το θέμα. Και έχουμε ένα νέο τρόπο σκέψης για την δημοσιονομική στήριξη. Η δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να είναι το συμβολέου χρηστή διακυβέρνηση. Είτε είναι τομεακή είτε είναι παγκόσμια, θα πρέπει να συναρτάται από όρου. Και η ισότητα των φύλων θα πρέπει να είναι ένα από του όρου αυτού που θα κρίνουν την αιρεσιμότητα τέτοιων συμφωνιών. Επίσης, θέλουμε απτά αποτελέσματα από τη συζήτηση με πλήρη εξοπλισμό όλων των αντιπροσωπιών και μάλιστα μέχρι το υψηλότερο επίπεδο και επίσης να υπάρχει λογοδοσία και να περιλαμβάνονται τη διάσταση των φύλων σε όλες τις πολιτικές τους. Και ευχαριστώ κυρία Φερνά για την παρατήρησή σας ότι δεν δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο θέμα ανάπτυξης. Είναι κάτι που ξεπερνά την ανάπτυξη. Ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις εξωτερικές ε, υπηρεσίες ε, και να αξιοποιήσουμε το καλό έργο που ήδη έγινε για την ισότητα των φύλων, για τις γυναίκες σε σειράξεις. Και επίσης έχουμε αυτή, αυτό το σούπερ έτος που θα ολοκληρωθεί με την διάσκεψη κορυφής των Παρισίων για το κλίμα. Και για κάποιο λόγο οι γυναίκες, ε, τα κορίτσια και οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι ε, στα θέματα των θεομηνιών, των φυσικών καταστροφών που είναι όλο και πιο ανθρωπογενείς όσο περνάει ο καιρός. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και δεν θα πρέπει να τη χάσουμε σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Χιμένες ζήτησε το λόγο, η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ, ο κύριος Τσέλερ και ο κύριος Στίερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Ήταν μερικές κάπως απογοητευτικές, παρόλο που ήταν και ρεαλιστικές ταυτόχρονα. Ήταν απογοητευτικές γιατί μας ε, κατέδειξαν την έλλειψη των ε, διαθέσιμων στοιχείων και την αδυναμία ε, συγκρότησης στατιστικών πινάκων. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να προβούμε σε εμπεριστατωμένη μελέτη αυτού του υλικού. Δεν έχουμε τη δέωση ευαισθησία προς τα προβλήματα μεταξύ των δύο φύλων και στις διαφορές και διακρίσεις βάρος των γυναικών. Στο θέμα της έμφυλης βίας, της εξιστικής βίας, βλέπουμε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ των 28 χωρών, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε την έκθεση για τα, για τα θύματα εγκλημάτων και είχαμε και ένα κεφάλαιο για την ε, έμφυλη βία, για τη σεξιστική βία. Ε, οι ίδιες δεν χαρακτηρίζονται με τον ίδιο τρόπο ως σεξιστική βία, για παράδειγμα, σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν ακόμη και μεταξύ μας. Επίσης, ε, σήμερα το πρωί, το είπαμε στην Επιτροπή και πρόσφατα στη συνάντηση που είχαμε τις χώρες ΑΚΕ, μιλήσαμε εκτενώς τουλάχιστον ε, εμείς οι Ευρωπαίοι και ο κύριος Στάβορ και εγώ το θίξαμε το θέμα του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι θέμα ε, παιδείας μερικές φορές. Ε, μιλάμε για πολιτιστικές διαφορές, αλλά υπάρχουν και κόκκινες γραμμές που θα πρέπει να είναι σταθερές. Ε, οι ακροτηριασμοί γεννητικών οργάνων, για παράδειγμα, ή η καταναγκαστική γάμοι που δεν έχουν καμία σχέση με τους συνενετικούς γάμους. Δεν είναι το ίδιο ένας γάμος συνενετικός και ένας αναγκαστικός, ενώ σε μερικές χώρες το αντιμετωπίζουν ως κάτι φυσιολογικό. Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι την νομοθετική διαδικασία στις χώρες αυτές. Γιατί για τις χώρες αυτές ακόμη και η καταναγκαστική γάμη είναι νομότυπη. Οπότε είναι πολύ περίπλοκο για μας. Είπατε ότι δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις ή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Και εγώ θεωρώ ότι οι κυρώσεις είναι το ίστατο μέσο, το έσχατο μέσο. Αλλά καλό θα ήταν να χρηματοδοτούμε μόνο συγκεκριμένα προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη διάσταση των φύλων για παράδειγμα. Διαπαιδαγώγηση για να αποφεύγεται ο κροτηριασμό των γεννητικών οργάνων, γιατί εκεί δεν μπορούμε να την απαγοράψουμε. Να την απαγορεύσουμε. Λυπούμε, αλλά τα πηγαδάκια δημιουργούν ένα θόρυβο στην αίθουσα. Παρακαλώ τη συζητήσει σα εκτός αιθούση, γιατί η συνάδελφο προσπαθεί να μιλήσει και δεν την ακούμε. Κυρία Μπεσερίλ, συνεχίστε. Είναι θέμα διαπαιδαγώγηση. Είναι πραγματικά επέσχυντο, γιατί οι, γυναίκες, οι άνδρες υποχρεώνουν τις γυναίκες να το κάνουν και οι γυναίκες ε, υποβάλλονται σε αυτή την επέμβαση γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να παντρευτούν. Για μας είναι αδιανόητο, αλλά για αυτούς είναι κάτι φυσιολογικό. Οπότε θα πρέπει να δράσουμε σε επίπεδο διαπαιδαγώγησης, σε επίπεδο παιδείας. Διαπαιδαγώγηση των αγοριών και των κοριτσιών. Μερικές φορές στέλνουν στο σχολείο μόνο τα αγόρια, γιατί τα κορίτσια θα τα παντρέψουν νωρί. Οπότε δεν δίνουν στον κόπο να τα στείλουν στο σχολείο. Γιατί σκέφτονται προ τι. Άχρηστο θα του είναι για το μέλλον ε, το σχολείο. Μάλιστα και για το φαγητό προτιμούν να σητήσουν πρώτα το αγόρι παρά το κορίτσι. Το αγόρι έχει προτεραιότητα. Σε όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε επίπεδο διαπαιδαγώγησης ένα άλλο ζήτημα, το θέμα του βιασμού των κορισιών και των γυναικών. Ο βιασμός χρησιμοποιείται ως όπλο στις ε, σειράξεις. Σας ευχαριστώ κύριε Μπεσερίλ. Ο κύριος Τζέλερ, μετά ο κύριος Στίερ, η κυρία Λόλα και θα ολοκληρώσουμε γιατί πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Yeah. Μα μπορώ να συνεχίσω απευθείας μετά από αυτά που είπε η Να τα συνδέσω. Φυσικά τα καλύτερα προγράμματα δράσης, τα καλύτερα προγράμματα χρηματοδότησης, όλα αυτά μπορούμε να τα προγραμματίσουμε, μέτρα κτλ. Το ερώτημα είναι, έχουν κανένα αποτέλεσμα. Η κυρία Χαουτάλα είπε να τους υποβάλουν ηλεκτροσόκ. Ε, εμείς δεν χρειάζεται, εμείς έχουμε ευαισθητοποιηθεί. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα στην συνάντηση ΑΚΕ αλλά και στη συνάντηση το Δεκέμβρη στην Ολομέλεια όλες οι προτάσεις που κάναμε μέσω ψηφισμάτων για τα θέματα αυτά επειδή υπήρχαν ε, πολλές ε, επιδράσεις δεν ξέρω ποιες αλίπητα απορρίφθηκαν από συναδέλφους αλλά και γυναίκες συναδέλφους ορισμένες φορές Άρα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση αυτό για να συζητήσουμε για περαιτέρω μέτρα. Αυτό τους είπαμε. Πρέπει να είναι προϋπόθεση. Και μας απάντησαν έχετε ο καθένας τις παραδόσεις και δεν θα πουλήσουμε εμείς τις παραδόσεις μας. Έτσι μας είπαν. Άρα δεν είναι θέμα προγραμματισμού. Είναι πρόγραμμα, πρόβλημα εφαρμογής. Με τους εταίρους μας γιατί αυτοί πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά. Πρέπει πολλά να κάνουμε ακόμη. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τέρους αυτές τις χώρες που δεν είναι στο πλευρό των κυβερνήσεων και κάποιων ισχυρών. Πρέπει να βρούμε άλλες μεθόδους. Να φτάσουμε στην κοινωνία των πολιτών. Αν υπάρχει ας πούμε κάποιο κίνημα γυναικών σε αυτές τις χώρες με το οποίο να μπορούμε να συνεργαστούμε αυτό βέβαια θα είναι πολύ πιο δύσκολο και πιο δαπανηρό από το απλώς να επιδιώξουν να υπάρχουν δεσμευτικές συνθήκες. Θεωρώ λοιπόν ότι τουλάχιστον οι εκπρόσωποι των χωρών ΑΚΕ που είναι στη νησομερή συνέλευση πρέπει να θεωρούνται από τα πιο πεφωτισμένα άτομα στη χώρα τους. Και με αυτούς δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρο. Ντάβο και Λόλα Σάντσε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και τους ομιλητές. Ευχαριστώ. Καταρχάς, πρέπει να χειραφετηθούν οι γυναίκες για την ανάπτυξη. Πολύ περισσότερο. Έχουμε γκρίνει τόσα ψηφίσματα γι' αυτό. Τουλάχιστον ε, οι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή συμφωνούν επ' αυτού. Επίσης, ότι η προσέγγιση μας πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό προωθούμε. Πρέπει όμως να γίνει μια διάκριση. Τι είναι ανθρώπινο δικαίωμα και άλλο μπορεί να είναι πρακτικές που είναι νόμιμες αλλά διεθνώς δεν, θεωρείται, δεν θεωρούνται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, στου ΑΚΕ, στο Φίτζι, επιχειρήσαμε να περάσουμε ένα πολύ ρωμαλαία διατυπωμένο ψήφισμα που εγκρίθηκε από όλε τι πολιτικέ ομάδε, από την ευρωπαϊκή πλευρά, με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά και από την πλειοψηφία των εκπροσώπων ΑΚΕ, που λέει σαφέστατα ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, να απαγορευθούν η ε, καταναγκαστική γάμη, οι ακροτηριασμοί γεννητικών οργάνων κτλ. Σαφέστατες διατυπώσεις. Αλλά επίσης ήταν σαφές ότι για ορισμένες άλλες πρακτικές που μπορεί να είναι νόμιμες σε κάποιες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως οι αμβλώσεις, οι ε, γάμοι ε, μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ότι αυτά δεν είναι ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να θεωρούνται θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσέγγισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ανάπτυξης. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Είναι ουσιώδης αυτή. Και ήταν ουσιώδης για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα που επιτύχαμε στην ε, ισομερή συνέλευση. Καλά, κάποιοι διαφωνούν μαζί μου. Ελπίζω η Χάιντι να μην μου κάνει ηλεκτροσόκ, που διαφωνώ μαζί της για το θέμα της άμβλωσης. Νομίζω ότι υπάρχει μια σαφή διάκριση που πρέπει να την κάνουμε για να εστιάσουμε επί των θεμάτων που είναι τα πιο σημαντικά για, την, για το αναπτυξιακό θεματολόγιο που μπορούμε να προωθήσουμε και να τύχουν συνένεσης. Ευχαριστώ και τελευταία η Λόλα Σάντσε. Ευχαριστώ. Κάτι που ξεχνάμε και που είναι απευθείας επίθεση κατά των γυναικών είναι λιτότητα. Βεβαίω πολύ σοβαρή στην Ισπανία η φυσική βία. 53 γυναίκες σε ένα χρόνο δολοφονήθηκαν στην Ισπανία. Μία τη βδομάδα. Είναι φρικόδες. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο αόρατο και σιωπηλό. Οι περικοπές στις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες. Όταν γίνονται αυτές οι περικοπές, οι γυναίκες την πληρώνουν. Έχουν επιπλέον καθήκοντα που προηγουμένως τα έκαναν κρατικές υπηρεσίες είναι γυναίκες που δεν μπορούν να εργαστούν ή δεν μπορούν πια να εργαστούν για να κάνουν ε, τις ε, θεραπεύτρες, τις νοσοκόμες, τις ε, νηπιαγωγούς. Χρειάζονται λοιπόν κάποιες μίνιμουμ υπηρεσίες. Χωρίς ένα μίνιμουμ επίπεδου οικονομικού οι γυναίκες υφίστανται τον, τον φαλοκρατισμό των ανδρών. Η λιτότητα είναι φαλοκρατική. Αυτό είναι πραγματικότητα. Μπορεί να είναι αόρατο, μπορεί να είναι ισοπηλό, αλλά υπάρχει. Επαναλαμβάνω. Κανείς δεν το λέει αυτό. Μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών, πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αν δεν το λάβουμε υπόψη, ό,τι και να κάνουμε θα έχουμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Μια ταχύτητα για τους άνδρες και μια για τις γυναίκες που θα πρέπει να κάνουν τα καθήκοντα που θα πρέπει να κάνει το κράτος. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, αν έχουν συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Ένα λεπτό ο καθένας, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε το φθινόπωρο στο θέμα αυτό κατά τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης στην Ολομέλεια. Οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν περισσότερο προς τον Ζαν Λουί για το μέλλον παρά για την αξιολόγηση. Είχαμε μερικές για την αξιολόγηση, λίγες για την Concord. Τζον, εσύ πρώτα. Ευχαριστώ. Επιγραμματικά. Για το ηλεκτροσόκ συμφωνώ, αλλά όχι πολύ δυνατό. Είμαι κατά των βασανιστήριων. Λίγα βόλτ λοιπόν στο ηλεκτροσόκ παρακαλώ. Τώρα, για τα δικαιώματα και τους κοινωνικούς κανόνες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε κάποιες κοινωνικές κανόνες. Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θέλουμε μία μεταστροφή στον τρόπο σκέψης, μία αλλαγή στον τρόπο σκέψης, όχι μόνο δική μας θεσμική, σε επίπεδο εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε ποια είναι η αξία, ποιες κοινωνικές, ποιοι κοινωνικοί κανόνες βρίσκονται πίσω από αυτή, πίσω από κάποιες πρακτικές και μια προσέγγιση που θα στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά εννοείται αυτός είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε και συζήτηση και με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτά και ευχαριστώ. Σεσίλ. Θα ήθελα και εγώ να αναφέρω ότι Πολλές χώρες ε, προσυπόγραψαν υποχρεώσεις ε, σε πολλές συμφωνίες και υπάρχουν βασικές ρήτρες για την πρόσβαση στην ε, υγεία, στο δικαίωμα για ασφαλή έκτρωση όπου είναι νόμιμη. Πολλά από αυτά τα συζητούμε και στο διάλογο πολιτικής και θα πρέπει να τα συζητήσουμε με τους εταίρους. Σε ό,τι αφορά τους προόρους γάμους, τους καταναγκαστικούς γάμους, τα προγράμματα που επεξεργαζόμαστε θα πρέπει να περιλαμβάνουν προσεγγίσεις που θα αναμειγνύουν και τους άντρες, γιατί έτσι θα αλλάξει η νοοτροπία. Δεν αρκεί να αλλάξουμε μόνο τους κανόνες και την νομοθεσία. Και αυτό δεν θα πρέπει να αλλάξει μόνο για το σχέδιο δράσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό κοινοβουλευτικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει για το πρόγραμμα αναπτυξιακή συνεργασία και τον προγραμματισμό. Γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε να δοθούν τα επαρκή κονδύλια για την ισότητα των φύλων. Κα, καλώς μας υπογραμμίσατε το ρόλο μας σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικό έλεγχο θα πρέπει να διενεργήσουμε στο μηχανισμό της αναπτυξιακής συνεργασίας, στο DCI. Δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Ντάκμαρ, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπατε για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και να τη χρησιμοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών για να απαιτήσουμε λογοδοσία από τις κυβερνήσεις. Και αυτό στο πλαίσιο των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων, αλλά και η χρηματοδότηση προς τους φορείς κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντική για να μπορέσουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους σε εθνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη λιτότητα, αποκοινούμε τον Ζαν Λουιβίλ και κάποιους άλλους που είναι στην αίθουσα. Ετοιμαζόμαστε για τη νέα εμβληματική μας πρωτοβουλία για τη νέα Παγκόσμια Έκθεση Προόδου για το 2015-2016 για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων, των οικονομικών δικαιωμάτων των γυναικών. Και εκεί εξετάζουμε και τον αντίκτυπο της λιτότητας. Έχουμε αντλήσει πολλά ε, διδάγματα από πολλές περιοχές του κόσμου που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και στο βορρά και στο νότο. Σας παραπέμπω στην έκθεση αυτή που θα είναι πολύ σημαντική, μπορείτε να αντιλήσετε και εσείς έμπνευση και θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί και το μελλοντικό πλαίσιο για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους ε, και την σχετική έκθεση. Υπάρχουν πολλά καλά μέτρα, αλλά δεν τα θέτουμε σε έμπρακτη εφαρμογή. Έχουμε αποδείξεις, έχουμε αναλύσεις, θα πρέπει να είμαστε τολμηροί και να δώσουμε προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων και στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Και αυτό θα κάνει και το σχέδιο δράσης ε, για, για την ισότητα των φύλων, το GAP θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτή την αλλαγή του τρόπου σκέψης, την αλλαγή της νοοτροπίας. Μόνο έτσι θα ε, καταλήξουμε σε ρηξικέλευτα μέτρα με φιλοδοξία και τόλμη. Αυτά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους καλεσμένους μας. Μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για το μελλοντικό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων. Παρακαλώ σκεφτείτε σοβαρά τη μορφή του εγγράφου. Μην το κάνετε εσωτερικό έγγραφο εργασία που ουσιαστικά απαξιώνει το έγγραφο. Δώστε τη μορφή της ανακοίνωσης ε, για να έχουμε εκτενείς διαβουλεύσεις και αποσαφηνίστε και οριστικοποιήστε το χρονοδιάγραμμα. Γιατί είναι απαράδεκτη αυτή η ελληπής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα. Χωρίς χρονοδιάγραμμα πώς να εργαστούμε και εμείς σωστά. Παρακαλώ, περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες. Ε, πολύ καλές πληροφορίες αυτές που λάβαμε για το τι έγινε μέχρι τώρα, τι χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε και τι ε, θα συμβεί με τις επικείμενες ε, παγκόσμιες διασκέψεις κορυφής για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ. Okay, so now we're going to have... Ωραία. Τώρα θα μιλήσουμε για το ECOWAS, ε, την οικονομική συνεργασία των κρατών της Δυτικής Αφρικής. speakers come to the platform. Παρακαλώ τους ομιλητές να έρθουν στο Προεδρείο. Okay, colleagues, we're going to go straight on. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε ακόμη δύο θέματα στην ημερήσια ταξι. Α, νόμιζα ότι κατεβαίνει ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, να περάσουμε στο σημείο 15. Πολύ σημαντικό. Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να έχω από πίσω μου να μιλάνε. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Είναι η οικονομική εταιρική σχέση της Ένωσης με τις χώρες της ε, Δυτικής Αφρικής. Έχουμε εδώ τον κύριο Φιέλμπερ, Φιέλνερ, ο οποίος είναι ο εισηγητής. Εμείς θα δώσουμε γνωμοδότηση για το θέμα της εταιρικής σχέσης, της οικονομικής εταιρικής σχέσης με το ECOWAS. Έχουμε μία έκθεση λοιπόν για να θέσουμε το πλαίσιο και έχουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες που θα μας μιλήσουν γι' αυτό. Η δόκτωρ Εβίτα Σμίγκ από το Γερμανικό Ινστιτούτο για Υποθέσεις Διεθνούς Ασφάλειας ήρθε το Βερολίνο. Η Μαρίκα Λέρτς που ήταν στη γραμματεία μας και δουλεύει στο, στην υπηρεσία ερευνών του Κοινοβουλίου και αυτή συνέταξε την έκθεση που ζητήσαμε για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές στην συμφωνία μας αυτή με την Δυτική Αφρική σε σχέση με άλλες οικονομικές εταιρικές σχέσεις. Είναι η μελέτη που ζητήσαμε. Μετά είναι ο κύριος Everdian Brower από την οργάνωση Concord και τον κύριο Γιάγια Σάου που είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος ε, του ΕΚΟΒΑΣ. Να δώσω λοιπόν πρώτα απ' όλα το λόγο στην δόκτωρα Βίτα Σμίγκ για έξι λεπτά. Θα περιορίσουμε τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. είναι τιμή που μπορώ να σας κάνω μια αποτίμηση για το ΕΚΟΒΑΣ. Πέντε σημεία θα αναφέρω. Το πρώτο είναι είναι μια νέα προσέγγιση για να, για να συνδυάσουμε την φιλευθερωπή του εμπορίου με την ε, βιωσιμότητα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ΑΚΕ έχουν αυτές τις συμφωνίες Ήθελα να έχουν ε, ένα μέσο που θα ήταν συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ και θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει το σύστημα εμπορικών προτιμήσεων με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ χρειαζόταν ε, μια κάποια αμοιβαιότητα. Δηλαδή και οι χώρες ΑΚΕ έπρεπε να ανοίξουν τις αγορές τους σε έναν βαθμό. Και έχουν γίνει πολλά σχόλια γι' αυτό, γιατί υπήρχε φόβος ότι τα τοπικά προϊόντα των αναπτυσσομένων χωρών θα κινδύνευαν. Δύο σημεία σε σχέση με αυτό. Πρώτον, η θεωρητική αλλά και η ε, εμπειρική ανάλυση έχει δείξει ότι η απελευθέρωση, ε, η φιλελευθερωποίηση δεν αυξάνει την οικονομική ανάπτυξη. Δεύτερον, οι θεωρητικέ αλλά και συγκεκριμένε πρακτικέ αναλύσει έχουν δείξει ότι ο προστατευτισμό επίση δεν αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη. Πολύ σημαντικά αυτά τα δύο γιατί καταδεικνύουν ότι ο λόγος για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας βασίζεται, είναι πολλαπλός. Έχει να κάνει σε μια σειρά, με μια σειρά από παραμέτρους αν οι χώρες είναι ανταγωνιστικές. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ΑΚΕ ήθελαν μια νέα προσέγγιση. Η οικονομική εταιρική σχέση είπα προσπάθησε να αξιοποιήσει την ε, φιλελευθερωποίηση του εμπορίου για να ψηφιακούς στόχους. Είναι πολύ νέα προσέγγιση. Δεύτερον, μπορεί κανείς να εφαρμόσει κριτήρια για να αποτιμήσει εάν οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να προωθήσουν την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Έγραψα ένα σύντομο κείμενο, νομίζω ότι σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά, οπότε θα είμαι σύντομη. Φαίνεται ότι οι συμφωνίες ΕΠΑ μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη. Το πρώτο που χρειάζεται είναι πραγματική πρόσβαση στις αγορές για τις αναπτυσσόμενες χώρες και μη συμμετρική φιλελευθερωποίηση. Η Ένωση έχει ανοίξει εντελώς τις αγορές στις χώρες εκεί. Είναι μεγάλη αλλαγή με αυτά που είχαμε προηγουμένως ε, κατά την σύμβαση του ΛΟΜΕ. Έχουν πραγματική πρόσβαση στην αγορά. Οι χώρες ECOWAS ε, χρειάστηκε να κάνουν πολύ πιο περιορισμένη ψηφοθροπήση και υπάρχουν και ευέλικτε ε, ασφαλιστικές ρήτρε για τις αναπτυσσόμενε χώρες και για την περιοχή συνολικά που επιτρέπουν να προωθηθούν πολιτικές όπως για παράδειγμα η σε κατάσταση κλάδη ή οικολογικές ε, προδιαγραφές. Θα αναπτύσσω περισσότερο στο κείμενό μου. Τρίτον, λοιπόν, κριτήριο συμβάλλει στην περιφερειακή ενοποίηση αυτή η συμφωνία. Εδώ είναι λίγο αντιφατικά τα αποτελέσματα. Το γεγονό ότι υπήρξε διπραγμάτευση για την ΕΠΑ βοήθησε την ε, περιφερειακή ενοποίηση γιατί ε, σήμαινε ότι οι χώρες αυτές ε, εφάρμοσαν κοινό δασμολόγιο. Αλλά υπάρχει κάποιος έστω και μικρός κίνδυνος ότι κάποια προϊόντα της Ένωσης θα αντικαταστήσουν τοπικά προϊόντα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό πρέπει οι χώρες αυτές να φιλοθροπήσουν και μία έναντι της άλλης. Αυτό προβλέπεται. Αλλά θα πρέπει να φιλοθροπήσουν τις σχέσεις τους με την ευρύτερη Ευρωπαϊκή, ε, Αφρικανική Ήπειρο. Μόνο έτσι μπορεί να βοηθήσει αυτή η συμφωνία για μία ευρύτερη ελεύθερη αγορά. Πώς ελέγχουμε τώρα την εφαρμογή. Η φιλελευθερωποίηση του εμπορίου μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ε, μείωση της τοπικής παραγωγής. και η μείωση των δασμών μπορεί να μειώσει τα κρατικά έσοδα. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε τι γίνεται κατά την εφαρμογή των συμφωνιών. Αυτό το προβλέπει αυτή η ΕΠΑ. Έκτο κριτήριο. Η φλευθεροποίηση συνδυάζεται με αναπτυξιακή συνεργασία. Η αναπτυξιακή συνεργασία βοηθάει τις χώρες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ε, αξιοποιήσουν έτσι πλήρως τη συμφωνία. Τρίτη υπόθεση. Οι ε, ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτές τις συμφωνίες δεν είναι καλύτερες δυνατές, αλλά είναι καλύτερες από το τίποτα. Θα τα πούμε και αργότερα. Σε άλλες συμφωνίες υπάρχουν καλύτερες διατυπώσεις για κοινωνικά θέματα ή για ανθρώπινα δικαιώματα. Παράδειγμα, το, η έπαγια του Κάρι Φόρουμ. Όμως ε, διαπραγμάτευση σημαίνει συμβασμός. Και για τις αφρικανικές χώρες ήταν πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό μια συμφωνία ΕΠΑ να αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της σύμβασης Κοτονού και δημιουργεί ένα πλαίσιο για τακτικό διάλογο και διαβούλευση για το θέμα αυτό. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα γεωπολιτικό επιχείρημα, ιδιαίτερα στα πλαίσια της μειούμενης ε, οικονομικής και πολιτικής σημασίας της Ένωσης σε πολλές περιφέρειες του κόσμου ε, και συμμετοχής. Τώρα, πότε θα αρχίσει η εφαρμογή. Γίνονται και άλλες διαπραγματεύσεις όμως για το TTIP με το Βιετνάμ και τα λοιπά. Και γι' αυτό οι εμπορικές προτιμήσεις θα χάσουν σταδιακά την ε, σημασία τους θα μειωθεί η αξία των ε, προτιμήσεων. Άρα είναι σημαντικό η εφαρμογή να αρχίσει σύντομα. Άλλο στοιχείο. Πέμπτο και τελευταίο στοιχείο συγκεκριμένα. Δεν είναι εγγυημένε οι θετικέ επιπτώσει αυτή τη και δεν είναι αυτονόητε και αυτόματε. Θεωρώ ότι η συμφωνία έχει ε, πρόπτικες. γιατί υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί δυναμικού που περιορίζουν τις δυνατότητες να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργεί η συμφωνία. Δεύτερον, μπορεί να υπάρχουν λόγοι πολιτικοί-οικονομικοί που μπορεί να εμποδίσουν τις αναγκαίες συνοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτός ο κίνδυνος ε, αφορά ιδιαίτερα την περιφερειακή φιλελευθερωποίηση, αλλά και για παράδειγμα τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να συνοδεύσουν αυτήν την μείωση των δασμών. Και αυτά που είδαμε από την ΕΠΑ του Κάρι Φόρουμ καταδεικνύουν το ΕΠΑ είναι μόνο ένα πλαίσιο. Άρα οι φορείς, ε, οι θεσμοί, αυτοί που εφαρμόζουν θα παίξουν τον ε, βασικό ρόλο για το πώς θα λειτουργήσει. Αυτή είναι η πρόκληση για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. I move now to um, Marieke Lurch, who has... Και τώρα θα Πρέπει να έχετε τη μελέτη αυτή, συνάδελφοι. Πρόκειται για μια μελέτη την οποία προετοίμασε το Τμήμα Πολιτικής και που εξετάζει τις ΕΠΑ της Δυτικής Αφρικής και τη συγκρίνει με άλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπόθηκε ότι ναι, το κείμενο αυτό πρέπει να το έχετε. Έχει δημοσιευθεί και στο ίντερνετ και να τονίσω ότι είναι πολύ τα δική μου ευθύνη αυτές οι θέσεις. Δεν είναι θέσεις επίσημες του Ευρωκοινοβουλίου. Θα συνοψίσω μόνο τα κύρια πορίσματα αυτής της μελέτης γιατί εκεί συμπεριλαμβάνεται και ένα μακρύ τεχνικό παράρτημα αλλά να πω και κάποιες πληροφορίες ε, όσον αφορά τους περιορισμούς μιας τέτοιας ε, ε, σύγκρισης. Καταρχήν το πεδίο της σύγκρισης ήταν περιορισμένο γιατί είχαμε μόνο μία ΕΠΑ ε, που μόλις αναφέρθηκε. Έχουμε μια διάμεση ΕΠΑ, αυτή είναι ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Αφρική αλλά βέβαια έχουν κάπως διαφορετική φύση και άρα θα πρέπει η αυτή, τη σύγκριση αυτή να τη δείτε πολύ προσεκτικά. Έπειτα ε, εστιάζουμε στις νομικές προβλέψεις και όχι στα, στις επιπτώσεις τους επιτόπου. Και είναι πολύ νέα η συμφωνία του ΕΚΟΒΑΣ για να δούμε και να μετρήσουμε το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις των διαφόρων προβλέψεων και διατάξεων. Υπάρχουν και άλλες ε, ε, εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν ε, το περιβάλλον επιτόπου και αυτές θα μπορούσαμε να τις αξιολογήσουμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Ακούσαμε σύντομα, ε, αν μπορέσουμε να συγκρίσουμε και τις τρεις ΕΠΑ, Διαπιστώνουμε ότι περιλαμβάνουν ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καλείται και ρήτρα μη εκτέλεση που εξασφαλίζεται μέσω σύνδεση με τη Σύμβαση του Κοτονού. Τα συμβαλόμενα μέρη μπορούν να προβούν σε κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το πλαίσιο ότι στη Συμφωνία του Κοτονού τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα ορίζονται μέσα στον ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλλον αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συμπεριλαμβάνει τις ε, προδιαγραφές ε, του Διεθνούς Οργανισμού Γραφείου. Ε, εργασίας, με συγχωρείτε. Έχουμε επίσης μια ε, αναφορά στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και στις τα καλύτερα περιβαλλοντικά ε, συμφέροντα και πρακτικές ε, που πράγματα που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε επίπεδο της εταιρικής σχέσης και έχουμε και κάποιες τομεακές προβλέψεις και διατάξεις στις τρεις συμφωνίες που αφορούν με την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα την γεωργία και την αλληλεία. Μουσική mm. Έχουμε εξετάσει συγκεκριμένα τις ΕΠΑ, ε, ε, περιλαμβάνουν και ένα κεφάλαιο για τα περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Είναι ένα ευρύ κεφάλαιο, προβλέπεται ότι τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νόμοι και οι πολιτικές που ακολουθούν θα προβλέπουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και θα πρέπει να συνεχίζονται, θα πρέπει να μειώνεται το επίπεδο προστασίας ώστε να επιτευχθεί ένα ανταγωνιστικό πλονέκτημα. Επιπλέον το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθησης και διαβούλευσης και εντός αυτών και τη δυνατότητα να ζητήσουν συμβουλές από τα αρμόδια διεθνή όργανα, ένας τρόπος δηλαδή να αποπολιτικοποιηθούν κάποιες διαφωνίες, καθώς και αν οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα μπορεί να συγκληθεί μια επιτροπή πυρογνωμόνων. Τώρα, κοινωνικές προδιαγραφές, ε, παρόμοια κατάσταση. Έχουμε κάποιες γενικές διατάξεις που αφορούν κοινωνικούς στόχους, κοινωνικές πολιτικές στην ΕΠΑ της Δυτικής Αφρικής και έχουμε και στις τρεις ΕΠΑ ρήτρες ασφαλείας που επιτρέπουν στις χώρες να μειώσουν τις ε, εισαγωγές αν υπάρχουν βασικά κοινωνικά προβλήματα. Ε, ε, για τις ε, εργασιακές ε, διαταξίες αυτές περιλαμβάνονται μόνο στην Συμφωνία Κάρι Φόρομα. Υπάρχουν δεσμεύσεις όσον αφορά το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, δέσμευση για τη τήρηση υψηλού επίπεδου κοινωνικών προδιαγραφών σύμμορφων προς τα διεθνείς προδιαγραφές εργασίας και επίσης υποχρέωση να μην επιτρέπεται η μείωση του επίπεδου προστασίας ε, προς χάριν πλεονεκτήματος ανταγωνιστικού. Και εδώ έχουμε προβλέψεις για ε, παρακολούθηση, όπως αυτή που προβλέπεται για τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και άλλη μια πτυχή ε, που συνοδεύει τη, στη συμφωνία Κάρι Φόρουμ, το πτυχή των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των κοινωνικών ζητημάτων είναι ότι περιλαμβάνεται μία διάταξη για την ρύθμιση των διαφορών και ως έσχατο μέσο όταν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ε, άλλες κυρώσεις δεν επιτρέπονται. Υπάρχουν δύο ακόμα κοινά στοιχεία που θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχήν και οι τρεις συμφωνίες πλαισιώνονται από την Συμφωνία του Κοτονού που περιλαμβάνει διατάξεις τα άρθρα 49 και 50 που αφορούν το περιβάλλον και τις κοινωνικές προδιαγραφές, κοινωνική πρόνοια, καθώς και εργατικά δικαιώματα τα οποία υπογραμμίζονται και υπάρχει και διάταξη για αύξηση συνεργασίας για αυτά τα θέματα. Όμως δεν υπάρχει διάταξη όπως υπάρχει στην Κάρι Φόρουμ για συγκεκριμένη διαδικασία παρακολούθησης ή διαβούλευσης. Ένα ακόμα κοινό στοιχείο που αφορά στις δύο περιφερειακές ε, ΕΠΑ, Κάριφορμ και Δυτική Αφρική, έχουμε θεσμικό πλαίσιο, ιδιαίτερα Κοινοβουλευτική Επιτροπή και Συμβουλευτική Επιτροπή που περιλαμβάνουν ε, κοινωνικούς και ε, οικονομικούς εταίρους καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Και αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι σημαντική γιατί ρητά αναφέρεται στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για θέματα περιβάλλοντος και ε, ε, για εργατικά θέματα. Έχουμε δηλαδή ένα θεσμικό πλαίσιο για διάλογο για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Συνοψίζοντας τώρα, τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά στι τρει συμφωνίε είναι η ρήτρα μη εκτέλεση που καλύπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, η, σύνδεση με, την Συμφωνία του Κοτονού και έπειτα ισχυρές διατάξεις όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα. Η βασική διαφορά είναι αυτά τα ειδικά ε, κεφάλαια που έχουμε στην ΕΠΑ Φόρουμ. Οι άλλε δύο θα πρέπει να βασίζονται σε αυτά που ήδη περιλαμβάνει η Σύμβαση του Κοτονού. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα. Και γι' αυτό οι ECOWAS και οι άλλοι για τη Δυτική Αφρική έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα του τι θα συμβεί όταν θα εκπνεύσει η Συμφωνία Κοτονού. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Με προλάβατε. Γιατί πριν από λίγο είχαμε πει κατά πόσο θα ανανεωθεί η Συμφωνία Κοτονού γιατί έχουμε πολλές εμπορικές συμφωνίες στο πλαίσιο της Κοτονού και δεν είναι βέβαιο το μέλλον της συμφωνίας Κοτονού, οπότε αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τι θα γίνει με τη συμφωνία Κοτονού και πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο μετά τη συμφωνία Κοτονού. Θα ακούσουμε τώρα πρόσωπο της ε, μη κυβερνητικής οργάνωσης Concord, τον κύριο Εύα Βαμπρόερ και μετά έναν εκπρόσωπο δυτικο, χώρο. Κύριε Μπρόιερ, είστε από το Ολλανδικό Ίδρυμα Word and Dad. Δεν το γνωρίζω, θα μας το περιγράψετε εσείς. τους του συμφωνίες ε, συμβάλλουν τελικά στην ανάπτυξη. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον για μας. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τις θέσεις της Concord ε, εκπροσωπούμε ένα ευρύ φάσμα διαπραγματε... Ε, οργανώσεων στην Concord. Το θέμα είναι κατά πόσο η ΕΠΑ, οι Συμφωνίε Οικονομική και Εταιρική Σχέση, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των χωρών τη Δυτικής Αφρική. Έχουμε εκπονήσει μία μελέτη σχετικά. Μάλιστα υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής σας. Μπορείτε να τη διαβάσετε. Θα σταθώ σε μερικά σημεία αυτής της έκθεσης. Η κοινωνία των πολιτών στις δικοαφρικανικές χώρες, ε, δυστυχώς δεν έχουν στείλει εκπροσώπους εδώ, ε, αγρότες, ε, συνδικάτα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, εκκλησίες, ε, ιδιωτικές ε, οργανώσεις, ιδιωτικός κλάδος της Δυτικής Αφρικής. Όλες αυτές οι οργανώσεις έχουν εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στη Δυτική Αφρική. Μερικές ήταν και ενάντια στην ΕΠΑ. Η Concord, η οργάνωσή μας έχει στενές σχέσεις ε, με τους συμμάχους μας ε, στη Δυτική Αφρική, τους εταίρους μας ε, στη Δυτική Αφρική και προσπαθούμε να διαμηνήσουμε τις ανησυχίες τους στους πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους νομοθέτες. Βέβαια, αν ήταν εδώ οι ίδιες οι οργανώσεις θα εξέφεραν καλύτερα τη θέση τους. Τώρα, για την ίδια την ΕΠΑ, την Συμφωνία Οικονομικής και Εταιρικής Σχέσης. Η πρώτη μελέτη επιπτώσεων που έγινε το 2004 για την ΕΠΑ για το τι μορφή θα πρέπει να έχει μια ιδανική ΕΠΑ, λέει τα εξή. Η ιδανική ΕΠΑ θα πρέπει να έχει τα εξή χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερων μεταποιημένων προϊόντων της Δυτικής Αφρικής και θα πρέπει να περιορίσει την πρόσβαση ε, ευρωπαϊκών προϊόντων σε χώρες Δυτικής Αφρικής εφόσον τέτοια προϊόντα μπορούν να παραχθούν και τοπικώς και επίσης θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για, μια, για εύρυθμες ε, περιφερειακές αγορές. Η περιφερειακή ολοκλήρωση θα, πρέπει να ενθαρρύνεται με την το, εγχώρια παραγωγή και την αξία της για τις ε, ε, περιφερειακές αγορές και τις αγορές προς εξαγωγή. Αυτό λέει η αξιολόγηση του 2004. Τώρα έχουμε, περάσει 11 χρόνια. Η παρατήρηση της Concord είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση στη Δυτική Αφρική. 13 από τις 16 χώρες που είναι εταίροι της ΕΠΑ ΕΚΟΒΑΣ έχουν ε, εμπορικό έλλειμμα και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και παρόλο που έχει αυξηθεί το εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Δυτικής Αφρικής 13 από τις 16 χώρες ε, αντιμετωπίζουν εμπορικό έλλειμμα. Επίση, επίσης, ό,τι αφορά το ακαθάριστο εχώριο προϊόν των χωρών αυτών το ΑΕΠ της Νιγηρίας ε, είναι περίπου 520 ε, δισεκατομμύρια, ενώ της Ολλανδίας είναι κατά 60% υψηλότερο. Και μάλιστα αν πάρουμε τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία, είναι 3.360 δισεκατομμύρια, ενώ της Λιβερίας είναι 1,95 δισεκατομμύρια. Οπότε ε, η γερμανική οικονομία είναι 1.900 φορές μεγαλύτερη από τη Λιβεριανή. Δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δυτικής Αφρικής και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη στις μεταξύ μας συμφωνίες. Τώρα, ποια είναι τα... οι βασικές ανησυχίες της Concord για τη συγκεκριμένη συμφωνία οικονομικής ε, εταιρικής σχέσης. Η πρώτη μας ανησυχία αφορά την ανταγωνιστικότητα παρόλο που ένα τμήμα των προϊόντων έχει αποκλειστεί, τα ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα, το 75% του εμπορικού όγκου παρόλα αυτά θα πρέπει να, ε, απελευθερωθεί. Και 11 χρόνια μετά την πρώτη αξιολόγηση, την πρώτη μελέτη επιπτώσεων, ε, δεν έχουμε τα βασικά στοιχεία για για τα αποτελέσματα στην παρούσα κατάσταση. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου εκπονεί μια νέα μελέτη και περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτή τη μελέτη και τι δείχνουν για τον αντίκτυπο στι αναπτυσσόμενες χώρε τη Δυτικής Αφρική αυτή τη ΕΠΑ. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν είναι για μα η βασική ανησυχία σε ό,τι αφορά την ΕΠΑ στη Δυτική Αφρική. Επίση, θα πρέπει να έχει δοθεί προτεραιότητα σε ισχυρά προγράμματα περιφερειακής ολοκλήρωσης γιατί κατάλαβα καλά αυτά που είπε η δόκτωρα Βίτα Σμιτ, Σμικ, είπε ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση στη Δυτική Αφρική θα πρέπει να είναι ταχύτερη από την ολοκλήρωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικής Αφρικής. Η εσωτερική περιφερειακή ολοκλήρωση θα πρέπει να είναι ισχυρότερη. Επίσης έχουν χαθεί πολλά εισοδήματα από τους δασμούς. Επίση, έχουν λάβει χώρα φορολογικές μεταρρυθμίσεις, διεύρυνση της φορολογικής βάσης, και παρά τη βελτίωση του φορεσπρακτικού μηχανισμού, οι χώρες αυτές εξαρτώνται από εμπορικούς δασμούς που θα καταργηθούν. Οπότε θα έχουν απώλεια τέτοιων εσόδων από τους δασμούς. Στην Ιγυρία, για παράδειγμα, θα χαθούν 30% των δασμολογικών εισοδημάτων ετησίως σε σχέση με μια μελέτη του 2013 που έκανε η Επιτροπή ΕΚΟΒΑΣ ε, ΟΟΜΑ. Τρίτη ανησυχία αφορά το χώρο πολιτικής θα περιοριστεί αυτός ο χώρος ε, της πολιτικής. Αναφέρθηκα ήδη στις εισαγωγικούς δασμούς, αλλά και στους εξαγωγικούς ε, φόρους, που είναι περισσότεροι από τις απαιτήσει του ΠΟΕ. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα του χώρου πολιτικής που θα συρρικνωθεί εξαιτία της ε, Συμφωνίας Οικονομικής και Εταιρικής Σχέσης. Αυτή είναι η βασική προβληματισμή και ανησυχία της Κονκόρντος προς τη Νέα ΕΠΑ. Επίση ίσως είναι υπερβολικέ οι απαιτήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Δυτική Αφρική. Κάποια στιγμή η, είπε, η Δυτική Αφρική το 60% απελευθέρωση θα ήταν ε, αποδεκτό, αλλά δεν το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τελικό συμπέρασμα ήταν 75% απελευθέρωση. Τέλος. Να σας παραθέσω εδώ μία νέα μελέτη της, του, Γενικού, του Ολλανδικού Συμβουλευτικού, της Ολλανδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία του Κοτονού και να κάνω και μερικές παρατηρήσεις για το περιεχόμενο της, των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης και τη διαδικασία του. Τα τελευταία χρόνια διαπραγματεύσεις είχαν στόχο την ε, ολοκλήρωση των ΕΠΑ με επικέντρωση στην ε, εμπορική πειθαρχία. Οι ΕΠΑ έχουν γίνει αυτοσκοπός αντί να συμβάλλουν στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της ε, Σύμβασης Κοτονού. Ένα άλλο σημείο της μελέτης λέει ότι στην οικονομική συνεργασία και το εμπόριο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνοχής. Η ευρωπαϊκή στρατηγική έχει στηριχθεί αμυγό σε μια εμπορική πολιτική, αντί να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη εμπορική και αναπτυξιακή πολιτική. Αυτά ήταν βασικά αίτια των προβλημάτων στη διαδικασία διαπραγμάτευση των ΕΠΑ το παρόν σύστημα προσωρινών ΕΠΑ ήταν ουσιαστικά μια επιβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, ε, δυτικοαφρικανικές χώρες. Τα αποτελέσματα δεν είναι αρκετά θετικά και οι νέες ενδείξεις για, μια, για ένα νέο εμπορικό συζύγιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυτικοαφρικανικών χωρών δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, και αυτό απηχεί την θέση πολλών εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών της Δυτικής Αφρικής. Ε, θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε ε, να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή που είναι η καθήλια αρμόδια για τις συμφωνίες αυτές οι οικονομικές εταιρικής σχέσεις, ότι η παρούσα εταιρική σχέση δεν συνάδει με τους στόχους της βιώσιμης ε, ανάπτυξης της περιοχής της Δυτικής Αφρικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, τελευταίος ομιλητής ο κύριος Γιάγια Σό, που είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος ΕΚΟΒΑΣ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την άποψή σας λοιπόν για αυτό το κείμενο. Δεν έχει επικυρωθεί έτσι, δεν είναι ακόμη από όλε ε, τις χώρες ΕΚΟΒΑΣ. Πείτε μας πώς έχει προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και χαιρετίζω την παρουσία εδώ και εκπροσώπων κάποιων χωρών της περιοχής. Βλέπω εδώ εκπρόσωπο της ε, ακτής Λεφαντοστού και εκπροσώπους του Μπενίν και του Τογκό. Η ακτή Λεφαντοστού έχει υπογράψει την ενδιάμεση συμφωνία από ό,τι ξέρω. να σας πω πώς εκτιμούμε αυτή τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την Ένωση. Η Δυτική Αφρική αποτελείται από 12 φτωχές ε, χώρες και 4 χώρες μέσου εισοδήματος. Η συμφωνία αυτή τη χάνει συνένεση στην στην ε, Δυτική Αφρική. Σε τρία βασικά θέματα. Η πρόσβαση στην αγορά, η ανάπτυξη και η πρόσβαση για τα προϊόντα μας στις αγορές. Ακόμη δεν έχουμε διαπραγματευτεί το εμπόριο υπηρεσιών. Κάπου έχω ακούσει να λέγεται ότι έχουν φιλελευθερωποιηθεί και οι υπηρεσίες. Ούτε καν δεν έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Οι υπηρεσίες ε, θα συζητηθούν αργότερα. Επιμένω ότι η προσέγγιση μας ήταν να συμμετέχουν όλοι, όλα τα κράτη, οι δημόσιες διοικήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια, τα περιφερειακά κοινοβούλια, καθώς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, δηλαδή ο ιδιωτικό τομέα και η κοινωνία των πολιτών. Επιμένω πάρα πολύ, η κοινωνία των πολιτών. Οι ενός παραγωγών και οι πανεπιστημιακοί. Όλοι συμμετείχαν. Και φυσικά και η Επιτροπή της ε, η Επιτροπή Ανάπτυξης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η ΟΜΑ. Θέλαμε λοιπόν να συμμετάσχουν όλοι. Και έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορούσαμε να έχουμε τις γνώμες όλων των φορέων και συγκεκριμένα των φορέων ε, της κοινωνίας των πολιτών, ε, των ενώσεων παραγωγών, και του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό δημιούργησε ε, ευρεία συνένεση σε επίπεδο υπουργών, υπουργικών συμβουλίων, κυβερνήσεων, αρχικών κρατών και όταν υπήρχαν σημεία όπου οι διαπραγματεύσεις ε, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν ορίστηκε ο πρόεδρος Μακεσάτης της Σενεγάλης για να βοηθήσει Έτσι καταλήξαμε σε μια συμφωνία που είναι εμπορική. Είναι συμφωνία ελευθέρου, ελευθέρων συναλλαγών αλλά έχει μια πολύ ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση γιατί θέλει να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα που είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και επίσης ε, θέλει να βελτιωθεί η δυνατότητα όλοι οι να λαμβάνουν αποφάσεις και ε, αντισταθμίσεις αν χαθούν φορολογικά έσοδα και επίσης θέλει να υπάρχει ειδική και διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των διαφόρων κλάδων. Πολλά θέματα, μια δεκάδα λοιπόν αφορά, θα ε, αναφέρω μερικά. Πρώτα απ' όλα εμπορική εταιρική σχέση όπου τονίζεται ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να περιέχει την πλευρά της φιλευθερωπής του εμπορίου αλλά να τη συνδυάζει με την ανάπτυξη. Υπόθηκε και αυτό. Βιώσιμη ανάπτυξη η οποία πρέπει να βασιστεί στην ε, αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Πολύ σημαντικό αυτό. Ένα άλλο θέμα η βιωσιμότητα της συμφωνίας EPA, EPA που βασίζεται στην ε, τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια και στήριξη για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Και έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης που λέγεται PAPET. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε για τη διαφορά που, τις διαφορές μάλλον που έχει αυτή η συμφωνία ECOWAS με τη συμφωνία κάρι Forum που μοιάζει να είναι πιο προωθημένη. Αλλά θέλω να πω ότι ο μηχανισμός για την επίλυση διαφορών που προβλέπεται στη συμφωνία αποδίδει πολύ σημασία στη διαβούλευση και την διαιτησία και προβλέπει τη συνεργασία και στον τομέα της ε, νομικής βοήθειας για τις χώρες μας σε περίπτωση ε, διανέξεων. Και υπάρχει δυνατότητα να προσφύγουμε και στους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Ήδη υπόθηκε ότι συμφωνούμε να ανοίξουν οι αγορές μας κατά 75% μέσα σε μία εικοσαετία και επίσης υπήρξε συμφωνία και για τους δασμούς. Επίσης υπάρχουν και μηχανισμοί προστασίας εμπορικών ε, συμφερόντων, anti-dumping. Και επίσης συμφωνία των ε, κλάδων που είναι σε εμβριακή κατάσταση. Δεν ξεχάσαμε λοιπόν ε, την ανάγκη ανάπτυξη διαφόρων κλάδων. Και επίσης υπάρχει και μια διάταξη που απαγορεύει σε ένα κράτος ε, την εξαγωγή προϊόντων προς άλλο κράτος όπου απαγορεύονται. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ως αποτέλεσμα οι συμφωνίες αυτές να έχουν ιδιαίτερα αναπτυξιακό χαρακτήρα και επίσης επιμείναμε στη συμμετοχή όλων στην εφαρμογή και ιδιαίτερα όλα αυτά τα κοινά όργανα διαχείρισης της Συμφωνίας ΕΠΑ σε όλα αυτά τα κοινά όργανα συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να πω όμως ότι μία από τις προκλήσεις που δημιουργεί η συμφωνία αυτή EPA είναι εάν θα υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση της αναπτυξιακής διάστασης. Το πρόγραμμα ΠΑΠΕΤ είναι το μέσο που θα μας επιτρέψει να καταστεί βιώσιμη συμφωνία. Να έχουμε δηλαδή έντονη ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας, οικονομιών μας και των εξαγωγών μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αύξηση των επενδύσεων. Για να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία πρέπει να υπάρξουν επαρκείς πόροι. Τα προγράμματα που θέλουμε να προωθήσουμε κατά προτεραιότητα πρέπει να τύχουν επαρκούς χρηματοδοτήσεως ούτως ώστε να βελτιώσουμε και να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Καταλήγοντας, καταλήγοντας. Χωρίς αυτή τη συμφωνία θα είχαμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να υπήρχε τρομερός κατακαιρματισμός της περιοχής ενώ η περιοχή μας ήταν πρωτοπόρα στην ε, εμπορική συνεργασία. Θα υπήρχε πραγματικά κατακαιρματισμός λόγω της επικάλυψης διαφορετικών ε, συστημάτων εμπορικών. Επίσης υπήρχε πρόβλημα λόγω του ότι η Γκάνα και το και αξί του ελεφαντοστού είχαν πρόβλημα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την ανταγωνιστικότητά τους διότι εξήγαν ήδη μέγα μέρος της παραγωγής τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είχαμε λοιπόν διαπραγματευτεί μια περιφερειακή συμφωνία κατά 60%. Αν φτάσουμε σε ένα ποσοστό 60%, ορισμένες χώρες δεν μπορούν να απελευθερωποιήσουν παρά μόνο 10 με 15% και αυτό δεν είναι βιώσιμο ούτε και επιθυμητό. Καμία χώρα της Δυτικής Αφρικής το κάνει αυτό. Μίλησα για τις υπηρεσίες πριν από λίγο, τώρα ο Μπερνάρ μίλησε για <laughs> τις ε, τελωνιακές, τα τελωνιακά έσοδα της Νιγηρίας, ε, δεν ξέρω πού βρήκε αυτά τα στοιχεία, πάντως εμείς με διαφορετικό τρόπο υπολογίσαμε και φτάσαμε σε διαφορετικά νούμερα για τη συγκεκριμένη χώρα, την Νιγηρία. Τώρα, η απώλεια των τελωνιακών δασμών είναι κάτι το σχετικό, γιατί ξέρετε ήδη ότι στην περιφέρεια έχουμε χώρες με πολύ χαμηλή φορολογική πίεση. Αρκεί να γίνουν μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις και οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί το ποσοστό των εσόδων. Αυτά λοιπόν πάντως εμείς η ΣΕΝΤΕΑ της Δυτικής Αφρικής επιθυμεί να συνεχιστεί η ανάπτυξη και στηρίζουμε τη συμφωνία που έχουμε συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστώ. Okay. thank you very much for that. Um, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την εικόνα που μας δώσατε των διαπραγματεύσεων από τη δική σας άποψη και τώρα έχουμε τον κύριο Φέλλον που είναι εισηγητής. Θα σας δώσουμε το λόγο πρώτο. Βλέπετε τι ωραία που σας συμπεριφερόμαστε εδώ έτσι στην Επιτροπή. Επιτροπή. Μόνο το που έρχεστε σας δίνουμε το λόγο. Είστε πολύ ευπρόσδεκτος εδώ κύριε Φέλλον και μετά οι υπόλοιποι οι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις σοκολάτες, ε, για την γραμματεία. Θα εισάγουμε σοκολάτες. Θα προωθήσουμε τη συνοχή στη σοκολάτα σε ολόκληρο το κοινοβούλιο νομίζω. Πάντως ήμουν εδώ γιατί ήθελα να σας ακούσω, ήρθα γιατί ήθελα να σας ακούσω, γιατί ξέρω ότι έχουμε γνωμοδότηση και έγραφα και αλλά δεν αντιπροσωπεύονται πάντοτε όλες οι οπτικές γωνίες αυτά τα κείμενα. Θέλω να κάνω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι ίσως προς την Κομισιόν, γιατί όταν διαβάζω και άκουσα σε διάφορους τομείς ότι η σχέση ανάμεσα στην σύμβαση, με, με τη σύμβαση Κοτονού είναι το κλειδί εδώ, γιατί ακριβώς αυτή διατηρεί τις ε, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές εντός της συμφωνίας. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψη της Κομισιόν. Πώς βλέπει την εκπνοή της σύμβασης του, κοτόνου του Κοτονού. Γιατί έχω ακούσει πολλά και διάφορα, διάφορες απόψεις. Ορισμένοι λένε ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό, ενώ άλλοι λένε πως ίσως να υπάρξει πρόβλημα λόγω αυτού. Άρα σίγουρα η Κομισιόν έχει την δική της άποψη. Και έπειτα, ε, κάποια στοιχεία πραγματικά, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τα όσα άκουσα από την ΕΚΟΒΑΣ και την Κόνκορτ, ότι δηλαδή η κοινωνία των πολιτών συμμετείχαν ή δεν συμμετείχαν σε όλα αυτά. Γιατί από την ΕΚΟΒΑΣ ακούω το ένα που λέει ότι ε, που λέει ότι η κοινωνία των πολιτών είναι μαζί σας, ενώ οι φίλοι μας από την Comcord, από την Ολλανδία λένε όχι. Ενώ ή συμμετείχαν ή δεν συμμετείχαν. Δεν έχει και ναι και όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν είναι εδώ. Μπορεί να μας απαντήσει. Τώρα δεν έχουμε εδώ εκτό από την Κόμκορτ ε, κάποιον άλλον από την κοινωνία των πολιτών για να μα ε, πει τι συνέβη. Νόρμπερ Νόιζερ, είσαι ε, εισηγητή για τη γνωμοδότηση εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για όσα μας είπατε. Παρά το ότι αποκλίνουν κατά πολύ. Και το γεγονός ότι αποκλίνουν κατά πολύ είναι που κάνει πιο δύσκολο για μας να αποφασίσουμε. Θα ήθελα να μας πείτε Γιατί ορισμένοι δεν βασίστηκαν περισσότερο στα αποτελέσματα που επιτύχαμε στο Κάρι Φόρουμ. Γιατί εκεί επιτύχαμε καλά αποτελέσματα. Γιατί στο ECOWAS λοιπόν ε, δεν ε, αντιγράψαμε αυτά τα αποτελέσματα. Κάτι άλλο που με εκνευρίζει είναι αυτές οι αναφορές στο κοτονού. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με το κοτονού. Κανείς δεν ξέρει πότε θα συμφωνηθεί, θα καταλήξει επιτέλους η συμφωνία με το ECOWAS. Τι έννοια έχει να αναφερόμεθα στο κοτονού, εφόσον δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Επίσης, έχουν υπάρξει επικρίσεις ότι δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη η κοινωνική και η περιβαλλοντική διάσταση και η συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών. Νομίζω ότι ήταν επαρκής. Η εκπρόσωπη με το ECOWAS είπε ότι θα δημιουργηθούν οι αναγκαίοι φορείς ούτως ώστε αργότερα να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών μου φαίνεται λιγάκι αυτό απόδειξε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμμετάσχει επαρκώς ή και καθόλου η κοινωνία των πολιτών. Αυτά είναι τα θέματα που θέλω να θέσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζέλερ, ε, σκιώδης ηγητής και μετά η Μαρία Χόιλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες που είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Από τον εκπρόσωπο ΕΚΟΒΑΣ είδα ότι είναι ιδιαίτερα υπέρ της συμφωνίας. Αλλά ποιον να πιστέψουμε, αυτόν που εκπροσωπεί αυτές τις χώρες ή την δημόσια γερμανική τηλεόραση η οποία την προηγούμενη Κυριακή στο περιοδικό που έχει για διεθνή θέματα είπε ότι τα αφρικανικά κράτη άλλη μια φορά μας εκβιάζουν, είναι οι κακοί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων αυτών Και έδωσα ένα παράδειγμα από την ε, Ουγκάντα για την οποία θέλουμε να υπάρξει χωριστή συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και για την Κάνα η οποία ε, από το 2009 έχει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου αυτή τη στιγμή στέλνει η Γκάνα τα πουλερικά της ε, προς την συγγνώμη, αντίστροφα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει το ε, πλεόνασμα της παραγωγής της προς την Ουγκάντα και καταστρέφει τους τοπικούς παραγωγούς. Άρα έχουν τεθεί ερωτήματα. Έχουμε κάποιο χρόνο, μερικές μέρες, για να ασχοληθούμε με το θέμα. Και αν δεν υπάρξει ισχυρή δέσμευση από πλευράς των κρατών της Δυτικής Αφρικής και από τους οικονομικούς παράγοντες της περιοχής αυτής ότι θέλουν να υπάρξει συμφωνία, τότε θα έχουμε πολλές δυσχέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Χόιμποκ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για μένα. Άκουσα ότι θα έχουμε πολλά πλεονεκτήματα, αλλά θα ήθελα να ξέρω λίγο περισσότερο το πλαίσιο. Για παράδειγμα, Πώς γίνεται η μελέτη επιπτώσεων. Δεν υπάρχει καμία μελέτη αντικτύπου από ό,τι μου είπατε. Εάν είναι συμβατή αυτή η συμφωνία με τους αναπτυξιακούς στόχους για παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει εκ των υστέρων. Αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Τώρα για την πρόσβαση στην αγορά. Διαπραγματευόμεθα μεταξύ μίας από τις ε, πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και μίας από τις φτωχότερες. 12 από 16 χώρες είναι μεταξύ των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών. Αυτές οι χώρες έχουν τη δυνατότητα ήδη όλα τους τα προϊόντα εκτός από όπλα ε, χωρίς δασμούς να τα εξάγουν στην Ένωση. Γιατί χρειάζεται πλέον συμφωνία. Και τώρα για αυτό το επιπλέον το συζητήσιμο που θα τους δώσουν θα ανοίξουν κατά 75% την αγορά τους στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Πώς θα προστατευθούν τα τοπικά προϊόντα. Δεν καταλαβαίνω. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Με ανησυχεί. Σε αυτήν την Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΠΑ. Και ποιες είναι οι μακροχρόνιες ε, προοπτικές αναπτυξιακές. Εμείς εισάγουμε από αυτούς κυρίως ε, πρώτες ύλες, γεωργικές ή άλλες, ε, ξύλο, μπανάνες, κακάο, ε, φυτικά έλαια. Και αυτά είναι πρώτες ύλες που κατόπιν προστίθεται πολύ αξία μέσω της κατεργασίας του στην Ευρώπη. Πώς λοιπόν μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά. Αντίθετα εμείς ε, εξάγουμε κατεργασμένα προϊόντα όπου εμείς έχουμε την προστιθεμένη αξία είναι πολύ δυσχερής λοιπόν αυτή η κατάσταση. Και η πρόορη φιλελευθερωποίηση μέσω της ΙΠΑ, φιλελευθερωποίηση του εμπορίου, θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Θα έχουμε καλύτερη πρόσβαση ακόμη στις πρώτες του ύλε. Οπότε χώρες αυτές θα αποκλειστούν ακόμη περαιτέρω από δυνατότητες ε, προστιθέμενης αξίας επιτόπου. Άρα οι χώρες αυτές ε, θα έχουν ακόμη πιο περιορισμένε δυνατότητες να αναπτύξουν την οικονομία τους, να προστατεύσουν την παραγωγή τους, να αναπτυχθούν. Και υπόθηκε ακόμη, νομίζω και πρόσωπος ε, του ECOWAS είπε θα μειωθούν και οι φόροι. Θα μειωθούν οι προπολογισμοί λοιπόν των κρατών αυτών. Και αυτό νομίζω ότι θα τις δυσχεράνε ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε και με απασχολεί ιδιαίτερα η γεωργία. Είναι ο κύριος τομέας της οικονομίας. 60% των απασχολουμένων, 80% των τροφίμων που καταναλώνουν είναι από την περιοχή τους. Εάν η συμπεριφορά της, αν σκεφτώ τη συμπεριφορά μας εμάς ως κοινή γεωργικής πολιτικής, έχω πολλές ανησυχίες. Αυτά που χρειάζονται είναι ήδη φιλελευθερωποιημένα. Έχουμε το παράδειγμα του γάλακτος. Εγώ είμαι παραγωγός γάλακτος. Έχουν μειωθεί οι ποσοστώσει ε, στην Ευρώπη. Έχουν μειωθεί οι γαλακτοκομικές μας εγκαταστάσεις. Έτσι θα υπονομεύσουμε το μέλλον τους. Ήδη τους ε, εξάγουμε γάλα σε σκόνη που κατόπιν το κάνουν γάλα και κυκλοφορεί εκεί στις αγορές και καταστρέφει την τοπική παραγωγή και έχει τρομερέ επιπτώσει. Εδώ και 20 χρόνια με ε, αγανακτούσε τρομερά το γεγονός ότι εδώ στην Ευρώπη οι συνάδελφοι λαμβάνουν χαμηλές τιμές και στην Αφρική οι παραγωγοί καταστρέφονται. Και θα επιδεινώσουμε ακόμη την κατάσταση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις, πάρα πολλές αντιρρήσεις. Και γι' αυτό λοιπόν θα υποβάλω πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρεις ομιλητές, τέσσερις ομιλητές έχουμε ακόμη, το πολύ δύο λεπτά, γιατί έχουμε μείνει πίσω και έχουμε ακόμη ένα θέμα. Ο Ντάβορ Στίερ πρώτα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Πολλά ερωτηματικά ανακύπτουν και από την απάντηση όλων αυτών των ερωτήσεων θα κρυθεί αν θα δώσουμε τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δεν μπορούμε να ανοίξουμε όλα τα σημεία της διαπραγμάτευσης. Κύριε Σμίγκερ, ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες, αλλά μου άρεσε ιδιαίτερα η δική σας παρουσίαση και η μελέτη σας. Δεν μας παρουσιάσατε ένα ρόδινο τοπίο της ε, οικονομικής και εταιρικής σχέσης, αναλύσατε τα υπέρ και τα κατά αυτής. Ποιες θα είναι οι συνέπειες για την ε, ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής μιας αρνητικής ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιας καταψήφισης της ε, οικονομικής εταιρικής σχέσης. Διάβασα και το έγγραφο της Concord. Είπατε ότι οι ψηλόβαθμοι εξωματούχοι της ΕΚΟΒΑΣ ε, υπέγραψαν στις 30 Ιουνίου περιφερειακή ΕΠΑ των πιέσεων που δέχτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μας κύριε Σόι, Κόνκορντ κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για άσκηση πίεσης στην έκοβα αυτό. Ευχαριστώ. Ο Κριστιαν Πρέντα, η κυρία Σαρτζεντίνη και ο κύριος Περέιρα. Κρίστιαν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ε, προσκεκλημένους μας. Εγώ είχα ερωτήσει, ε, αλλά με πρόλαβαν οι συνάδελφοι. Τι γίνεται με το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Γιατί δεν κατάλαβα. Είχαν εμπλακεί οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών. Έγιναν διαβουλεύσει. Και τι σημαίνει ποσοτικά εσωτερική διαβούλευση. Έγινε καταρχήν και σε τι έκταση. Επίσης έχω την αίσθηση ότι δεν θα πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πέσουμε για μία ακόμη φορά στην παγίδα της αυτοκριτικής, της αυτομαστίγωσης που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι ε, όλων των δεινών. Και ότι εμείς είμαστε ακόμη και πιο υπεύθυνοι από τους ε, τοπικούς ε, πολιτικούς και τις τοπικές πολιτικές ελίτ. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να κάνουμε αυτή την αυτομαστίγωση, γιατί οι πρωταρχικές ευθύνες βαρύνουν τα καθεστώτα και τους πολιτικούς της περιοχής. Τέλος. Ανάγκη σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται και στο προήμιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης η δέσμευση των συμβαλωμένων μερών να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε παρόλα αυτά να λαμβάνουν χώρα ε, πολιτικές κρίσεις ε, και βλέπουν πόσο ευάλωτες είναι μερικές από τις χώρες αυτές. Τόσο ευάλωτες που δύσκολα μπορούν να τηρήσουν την υποχρέωσή τους για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να το αναλύσουμε εκ του σύνεγγης. Και να μην αυτοστιγματιζόμαστε και να διαρριγνύουμε τα μάτια μας ότι εμείς φταίμε περισσότερο από τους ε, πολιτικούς ε, και τις κυβερνήσεις των χώρων αυτών. Προσοχή. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις ε, διατυπώθηκαν και από τη Μαρία Χόιμπουργ. Θα τις αναπτύξω περαιτέρω. Άκουσα από τον εκπρόσωπο της ΕΚΟΒΑΣ ότι υπήρχαν χρονικές πιέσεις και κίνδυνος να επιδεινωθεί το εμπόριο. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα των διαπραγματευτών ε, σε διπλωματικό επίπεδο και όχι σε πολιτικό επίπεδο, γιατί οι αποφάσεις αυτές σε τελική ανάλυση έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Και η Δυτικοαφρικανική Ένωση ε, είπε ότι θα πρέπει ολόκληρη περιοχή να αντιμετωπιστεί ως ε, λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα οδηγήσει σε συμφωνία οικονομική εταιρική σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πρόθυμη να πάει στον ΠΟΕ και να ζητήσει ε, κάτι τέτοιο για τη Μολδαβία που είναι λιγότερο αναπτυγμένη χώρα στο ευρωπαϊκό έδος. Και αν ζητούμε εξαίρεση για τη Μόλδοβα, γιατί να μην ζητούμε εξαίρεση για την ΕΚΟΒΑΣ. Είναι πρόβλημα αυτό γιατί ξέρουμε πού θα μα οδηγήσουν όλα αυτά. Και ξέρουμε ότι δεν θα γίνει επαρκής διαβούλευση με τα ε, Εθνικά Κοινοβούλια. Ποτέ δεν γίνεται κάτι τέτοιο γιατί δεν υπάρχει νομική υποχρέωση. Αλλά το συζητούμε εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οδηγούμαστε σε μια παράδεκτη κατάσταση. Γιατί είναι σαν να γνωρίζουμε εμείς καλύτερα τα πράγματα από τις ε, δικοαφρικανικές χώρες. Αλλά εμείς ε, αφουγκραζόμαστε και τις δικές μας κοινωνίες των πολιτών που έχουν στενές επαφές με τις δικές τους κοινωνίες των πολιτών. Και πολύ θα ήθελα να έχουμε ε, εθνική συζήτηση ή ε, συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί μερικοί από σας πήγατε στο Φίτζι και είχατε συναντήσει με βουλευτές των χωρών ΑΚΕ. Και πολύ συχνά μας εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο διαπραγμάτευσης των συμφωνιών οικονομικής εταιρική σχέσης. Δικαιούμαστε λοιπόν απαντήσεις. Και δεν θα πρέπει να μας αρκεί το σχόλιο ότι είναι πατερναλιστικό να λέμε ότι η συμφωνία είναι κακή ο Πέδρο Σίλβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται πάντα σε δύσκολη θέση. Γιατί μετά από μια μακροχρόνια διαπραγματευτική διαδικασία καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι για το κατά πόσο μια συμφωνία είναι βιώσιμη. Πολλό δε μάλλον που η συμφωνία αυτή έχει γίνει με 16 άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να, να ληφθεί υπόψη και η δική τους γνώμη και η δική τους θέση. Διατυπώθηκαν πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Εγώ θα περιοριστώ σε δύο και να ζητήσω από τους καλεσμένους μας να μας βοηθήσουν για να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση. Για να είναι ευνοϊκή μια τέτοια συμφωνία στην ανάπτυξη, θα πρέπει να είναι πραγματικά ασύμετρη. Το είπαν οι πυρογνώμονες μας. Το θέμα είναι η συγκεκριμένη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης είναι όντως ασύμετρη. Ο βαθμός δηλαδή απελευθέρωσης ή φιλελευθεροποίηση του εμπορίου που απαιτείται από τις χώρες ΕΚΟΒΑΣ είναι βιώσιμη για τις οικονομίες τους, που είναι αναπτυσσόμενες οικονομίες και είναι αρκετά μακροχρόνια η μεταβατική περίοδος, είναι επαρκής. Αναφέρθηκε απώλεια φορολογικών εσόδων από τους δασμούς. Θα πρέπει να αντισταθμιστούν αυτές οι δασμολογικές απώλειες από προγράμματα συνεργασίας ή από άλλα αντίβαρα ή από άλλα αντισταθμιστικά ωφέλη. Εμείς σημειώνουμε ότι υπάρχουν προγράμματα συνεργασίας. Ερωτώ όμως και πάλι, αυτά τα εναλλακτικά έσοδα, αυτά τα αντισταθμιστικά ωφέλη επαρκούν για να αντισταθμίσουν την απώλεια των δασμολογικών εσόδων. Αυτά τα τεχνικά στοιχεία για την αξιολόγηση του αντικτύπου της συμφωνίας έχουν κέρια σημασία για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογήσει τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας ΕΠΑ. Μια άλλη σημαντική ερώτηση ήταν Ποιε θα είναι οι συνέπειες μιας απόρριψης της Συμφωνίας ΕΠΑ, Συμφωνία Οικονομική Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκοβα. Um, Σα ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο ε, στους ομιλητέ μας, έχω εδώ τρία ονόματα για την Κομισιόν. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει το λόγο. Κυρία Γκαλίνα από την ε, DG Trade, ο κύριος Κοκοτσίδης ή κάπως έτσι. Ε, πάντως δεν μπορώ να τα διαβάσω καλά. Κι άλλος ένας είστε από τη Digitrade πρώτα. Σύντομα παρακαλώ όμως. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους ε, επίση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε και θα απαντήσω στις λίγες ερωτήσεις που ε, ανέκυψαν στη διάρκεια του απογεύματος. Καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται γνήσια για μια αναπτυξιακή συμφωνία. Η ανάπτυξη δεν είναι ένα από τα στοιχεία της συμφωνίας και η συζήτηση που μόλις έγινε μου δείχνουν ότι ίσως θα ήταν καλό να κάνουμε και μια τεχνική συνεδρίαση που να σας αποδείξω γιατί πρόκειται για μια συμφωνία που πραγματικά υπερασπίζει την ανάπτυξη. Να τονίσω ότι έχουμε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για να συνοδεύσουμε αυτή την περιοχή όχι μόνο μέσω της απελευθέρωση αλλά και ακόμη περισσότερο και αυτό βρίσκεται μέσα στην συνθήκη στο άρθρο 54.3 Έχουμε μια ολόκληρη σειρά στοιχείων που ε, παρουσιάστηκαν, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, αλλά για τις απώλειες, τις ε, δημοσιονομικές απώλειες. Έχουμε το άρθρο 60 που έχουμε δέσμευση για να προωθήσουμε την προσαρμογή και να καλύψουμε τις απώλειες που προκύπτουν από αυτή τη συμφωνία. Και, ε, εδώ παραθέτω την πολύ πρόσφατη μας μελέτη από την Παγκόσμια Τράπεζα που λέει ότι η ΕΠΑ όπως είναι δομημένη τώρα γιατί οποιοδήποτε μελέτη αντικτύπου που είναι επεπαλαιωμένη κάνει δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Η Παγκόσμια Τράπεζα λοιπόν βλέπει την ΕΠΑ όπω είναι δομημένη και λέει ότι οι μεγάλε οικονομίε όπω η Νιγηρία η απώλεια στο τέλο της δικασία, 20 χρόνια μετά δηλαδή θα είναι 0,8% των εσόδων τη χώρα. Αυτό στο τέλο. Στι αρχέ είναι σχεδόν μηδενικέ οι απώλειε. Α κάνουμε λοιπόν μια τεχνική συνεδρίαση για αυτά τα ζητήματα αν θέλετε. Και κάποια άλλα θέματα. Η ε, φόροι εξαγωγών ε, και αυτοί περιλαμβάνονται εδώ. Δεν θέλω να ακούω καταγγελίες για δήθεν ε, απόλυση τέτοιο οι μη λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες τώρα ναι βεβαίως έχουν, έχουν περιφερειακή αντιμετώπιση αλλά υπάρχουν κανόνες προέλευσης που θα έλεγα είναι πολύ ευνοϊκοί, εξαιρετικά ευνοϊκοί είναι η οι κανόνες προέλευσης που έχουμε δώσει και για τους ε, ε, αδερφούς μας από την Ανατολική ε, Ευρώπη. Τώρα, για τα κοτόπουλα και το γάλα είναι αυτά παραμύθια. Είτε μπορείς να σταματήσεις τις ευρωπαϊκές εισαγωγές. Δεν είναι ευρωπαϊκές εισαγωγές. Τα περισσότερα από κοτόπουλα έρχονται από τη Βραζιλία. Και έπειτα, θεμελιώδη ερώτημα είναι στο δισκοτονού. Και εσείς, Πρόεδρε, είπατε και σωστά ότι αυτές οι συμφωνίες βασίζονται στην διαδικασία του Κοτονού και είναι πολύ σημαντικό που κάνετε αυτή τη δήλωση γιατί δείχνει ότι για μας το Κοτονού είναι πολύ σημαντικό τμήμα αυτής της συμφωνίας. Να πω επίσης ότι η Κοτονού είναι μια μνημειώδης δομή. Είπατε ότι έχουμε την παιδική εργασία, έχουμε τη διαφθορά, οποιοδήποτε θέμα περιλαμβάνεται και είναι μια καταπληκτική δομή αυτή η συμφωνία. Τώρα, εσείς ανησυχείτε και δικαίως ε, για την εκπνοή της το 2020. Καταρχήν επιτρέψατε μου να πω ότι κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να σεβόμαστε τα συμβαλόμενα μέρη ε, που σήμερα υπέγραψαν με αυτό το ιστορικό και δεν ευχαριστούνται όταν ακούνε κάποιον που να λέει ε, τι θα γίνει το 2020. Έχουμε λοιπόν την Συμφωνία του Κοτονού και νομικώς τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει μια επίπτωση που είναι κάπως λεπτή θα μπορούσα να πω και να σας πω ότι όταν θα εκπνεύσει η σύμβαση του Κοτανού θα έρθουμε και θα ξαναδιαπραγματευτούμε. Και αυτό είναι ε, εφικτό γιατί έχουμε σχετικές ε, ρυθμίσεις και ρήτες. Πάντως σήμερα ε, έχουμε μία συμφωνία, έχουμε συμφωνίες υπογεγραμμένες επί τη βάση αυτών των βασικών στοιχείων και μπορούμε να εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα επί τη βάση αυτών των, αυτής της συμφωνίας. Αυτές είναι οι νομικές ε, προσδοκίες, οι νόμιμες προσδοκίες, θα σας πει οποιοδήποτε καλός δικηγόρος και καλός νομικός, ότι ούτως ή άλλως εφόσον εκπνεύσει η Συμφωνία του Κοτονού, εμείς αυτά αναμένουμε από τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει. Έχουμε από κοινού συνυπογράψει, εν πάση περιπτώσει τώρα θα γίνει η κύρωση της συμφωνίας, δηλαδή μην το διωγγώνουμε ως πρόβλημα, γιατί βεβαίως το Κοτονού, εάν υπάρξει διάδοχη συμφωνία, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό γιατί όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές. αλλά εν πάση περιπτώσει η σημερινή συμφωνία υπογράφεται με τις ε, νόμιμες προσδοκίες ότι τα βασικά της στοιχεία της Κοτονού θα γίνουν σεβαστά. Έπειτα η συνθήκη Λισαβόνας 2.15, άρθρο 2.15 λέει ότι πάντοτε ε, πρέπει να σεβόμαστε τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και έχουμε ένα, μια ολόκληρη δηλαδή, ε, ένα ολόκληρο πλωστάσιο από μέσα για να στηρίξουμε αυτές τις συμφωνίες. Και έπειτα εφόσον είμαστε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, όπως είπε και ο δόκτωρ Σμίγκ, ότι έχουμε ένα στοιχείο το οποίο δυσκολεύει, ε, είναι η παρακολούθηση αυτών των συμφωνιών. Και εδώ σχεδόν έκκληση σα υποβάλλω. Σε αυτήν εδώ τη συμφωνία έχουμε κοινοβουλευτική συνέλευση και έχουμε και την κοινωνία των πολιτών και έχουμε και ένα παρατηρητήριο. Μπορείτε να μας βοηθήσετε στην παρακολούθηση. Εγώ βλέπω σημαντικό ρόλο για το Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση και την υποπτία, γιατί είναι ένα ε, τομέα όπου θα είχαμε αποδείξει. Οι συμφωνίε μπορεί να είναι καλέ ή κακές ε, στα χαρτιά και ειλικρινά εγώ είμαι περήφανη για αυτή τη συμφωνία γιατί οδηγεί σε πολιτική συνοχή με την πλήρη έννοια τη φράση αυτή, Έπειτα θα είναι καλή, όμω από την άλλη πλευρά επί τη βάση του τι, τι θα κάνουμε εμεί στην πράξη. Ζητώ συγγνώμη που καθυστερώ να δίνω το λόγο στον συνάδελφο. Θα ήθελα όμως ο συνάδελφος Ντιντιέ, ε, ε, γιατί η στήριξη για τη Γεωργία είναι πολύ, πολύ σημαντική. Μάλιστα, λέει πρόεδρος, όσο γίνεται πιο σύντομα. Βασική μας στοιχεία είναι η Έχετε κάνει εσείς την αξιολόγησή σας, τι έχετε να μας πείτε. Ναι, πολύ σύντομα λοιπόν. Για το τμήμα της, ε, το αναπτυξιακό υπάρχει ένα θέμα που δεν έχει προβλεφθεί, επιπλέον ταμεία. Ας μην τις φορτώσουμε με πλέον κονδύλια. Τώρα, όσον αφορά το 11ο ΦΕΔ, οι τομεί σε συγκέντρωση έχουν οριστεί σε συνοχή με τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε τον Ιανουάριο του 2014 απέναντι στις συμφωνίες ΣΕΝΤΕΟ και ΟΜΑ. Ε, δηλαδή, γεωργία, ενέργεια, μεταφορές, αλλά και περιφερειακή ολοκλήρωση και στήριξη στην κοινωνία των πολιτών που σαφώς αναφέρθηκε, έχουμε, ε, ε, έχουν προτεραιότητα στο 11ο ΦΕΔ. Αυτό έχει προβλεφθεί από το συνδευτικό πρόγραμμα. Υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Απριλίου του 2000, συγγνώμη, Μαρτίου 2014 5 δις ευρώ σε συνοδευτικά μέτρα. Συγγνώμη, 6,5 δις. 3 δις που θα προέρθουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 1 δις από την ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω υποδομών για τη Δυτική Αφρική και δύο δις θα προέλθουν από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τα τρία δις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα διάφορα μέσα, αλλά βασικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Αναπτυξιακό και το Γενικό ε, Ταμείο μέσω της ΕΝΤΕΟ και της ΟΜΑ, ε, ε, θα χρηματοδοτηθούν οι μικροί γεωργοί, αλλά και προγράμματα για την ενέργεια και τις μεταφορές μέσω της, ε, ε, ενός ε, μίξ χρηματοδότησης προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης έχει επηρεαστεί για να συνοδεύσει τις δυτικοαφρικανικές χώρες αυτό το εγχείρημα ανταγωνιστικότητας περιφερειακής ολοκλήρωσης και γεωργικής παραγωγής που είναι ο πρώτος τομέας ε, όπως γνωρίζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ε, τον, τους φορείς συγκέντρωση αλλά είναι και ο πρώτος οικονομικός φορέας της Δυτικής Αφρικής φυσικά και θα τους στηρίξουμε μέσα από τα διάφορα μας προγράμματα τα διμερή και τα περιφερειακά αλλά και τα θεματικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος ομιλητής. Ναι, παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος. Ο κύριος Σο πρώτα. Μάλιστα, πολύ σύντομα. Η κοινωνία των πολιτών συμμετείχε σε διάφορα επίπεδα στις διαπραγματεύσεις. Και το λέω και το επαναλαμβάνω συμμετείχε η κοινωνία των πολιτών στον καθορισμό της θέσης, της διαπραγματευτικής θέσης μάλλον, και σε κάθε συνεδρίαση διαπραγματευτική εκπροσωπούνταν στην αντιπροσωπεία κάθε χώρας και μιλώ για την Εθνική Κοινωνία των Πολιτών καταρχήν και έπειτα στην Επιτροπή των Διαπραγματεύσεων έχουμε και την Περιφερειακή Κοινωνία των Πολιτών. Είχαμε λοιπόν διαβουλεύσεις με όλα τα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα, Ας, ε, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Άκουσα λένε ότι η πρόσφορα, πρόσβαση στην αγορά δεν ήταν αρκετά καλή. Εγώ λέω όχι. Όταν λέμε ότι πρόκειται για άνοιγμα 75% είναι μια περιφερειακή συμφωνία. Δεν σημαίνει πως όλες οι χώρες θα απελευθερώσουν κατά 75%. Όχι. Είναι μέσο όρο. Α πούμε, η Γκάμπια μόνο 46%, το Μπενέν μόνο 58%. Άλλοι 64, ε, ε, άλλοι 70%. Είναι η ακτή του ελεφαντοστού που θα απελευθερώσει σε επίπεδο 81%. Αλλά ήδη είχε συμφωνήσει στην ενδιάμεση συμφωνία για να ανοίξει κατά 81%. Είναι μια, ένας μέσος όρος. Δεν σημαίνει ότι και η Γουινέα και το Μπενέν και το Μαλί και όλοι θα απελευθερώσουν σε επίπεδο 75%. Έπειτα έχουμε προστατεύσει όλα τα προϊόντα που προέρχονται από τη Γεωργία. Όλα και την κτηνοτροφία. Προστατεύθηκαν, δεν απελευθερώθηκαν και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έχουμε επίσης ε, φροντίσει για την αποζημίωση της καθαρής δημοσιονομικής επίπτωσης, για ε, την κάλυψη αυτής. Όπως το είπε και η Κομισιόν, έχουν γίνει συγκεκριμένες προσπάθειες όσον αφορά την ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, διαφοροποίηση της οικονομίας, υποδομές και επίσης ε, υπάρχει ε, παρακολούθηση της δημοσιονομικής προσπάθειας, ώστε η εξωτερική και εσωτερική ε, δημοσιονομική κατάσταση να εξισορροπηθεί και ίσως να έχουμε και δημοσιονομικό πλεόνασμα. Πάντως ε, δεν είναι σωστό να λέμε ότι οι προτιμησιακές ε, ε, αυτές συμφωνίες δεν προσέφεραν τίποτα στη Δυτική Αφρική. Διαφορετικά μπορεί να είχαμε καταρρεύσει, γιατί είχαμε διαφορετικά προτιμησιακά καθεστώτα. Εμείς είμαστε μια περιφερειακή ενότητα, προσπαθούμε να σας μοιάσουμε. Καταργήσαμε τις θεωρήσεις, τα τελωνία και σκοπεύουμε να φτιάξουμε και κοινωνόμισμα. Αν όμω, δεν δεχτείτε την ε, περιφερειακή ΕΠΑ, δεν θα τα καταφέρουμε. Η Ελληνική Ένωση θα αποσυνθεθεί και δεν θα υπάρξει αυτή η ε, ΣΕΔΟ. Και έχουμε διάφορα πρότυπα. Έχουμε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα έκαναν τις σχετικές εκθέσεις και τα βρήκαν όλα θετικά. να μην παρανοηθώ. Θεωρώ ότι είπα είναι θετικές. Είναι βέβαια διαφοροποιημένη προσέγγιση μου, αλλά δημιουργούν καλό κλίμα. Δημιουργούν καλές ευκαιρίες και έχουν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Και τα λέω περισσότερο στο έγγραφό μου. Η πρόσβαση των αγορών 100% είναι κάτι που δεν το δίνει στις χώρες Αφρικής καμία άλλη βιομηχανική χώρα και είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαν ε, υπό το κοτονού. Όπως είπε ο κύριος Σό, νομίζω ότι υπάρχει επαρκής ασυμμετρία, αλλά ούτως ή άλλως έχουμε το μηχανισμό παρακολούθησης. Και το Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Υπάρχει παρακολούθηση, υπάρχει επιτηρήση. Αν προκύψουν προβλήματα, υπάρχει η αναγκαία ευελιξία για να αντιμετωπιστούν. για την απώλεια ε, δημοσιονομικών εσόδων λόγω μείωση των δασμών. Αυτό θα είναι μακροπρόθεσμο. Θα γίνει μετά από 20 χρόνια, όταν θα υπάρξει αυτή η απελευθερωποίηση. Μόνο εάν το εμπόριο που έχουν αυτές οι χώρες θα είναι το ίδιο με αυτό που είναι τώρα. Και αν δεν υπάρξει φορολογική μεταρρύθμιση. Αλλά δεύτερον, η φορολογική μεταρρύθμιση είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη. Γιατί είναι πολύ κακό οι χώρες να εξαρτώνται από εισαγωγικούς δασμούς για τον προϋπολογισμό τους. Και αυτό επηρεάζει και την περιφερειακή ενοποίηση, διότι παρεμποδίζει την περιφερειακή ενοποίηση. Χρειάζεται λοιπόν φορολογική μεταρρύθμιση ούτως ή άλλως. Για τις επιπτώσεις ο κύριος Σόν νομίζω ότι τόνισε τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δεν υπάρξει συμφωνία θα δημιουργηθούν προβλήματα για την περιφερειακή ενοποίηση. Γιατί οι πιο ανεπτυγμένε χώρες χρειάζονται τη συμφωνία για να διατηρήσουν χρειάζονται την συμφωνία για να διατηρήσουν την πρόσβαση στις αγορές των άλλων χωρών. Δεν θα υπάρξουν λοιπόν περισσότερε ευκαιρίες αν δεν υπάρξει συμφωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ΕΠΑ αξίζει τον κόπο. Πρόεδρος, παρακαλώ. Εσείς κυρίως συλλέγετε στοιχεία έτσι δεν είναι ότι οι χώρες θεωρούν ότι θα υπάρξουν μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα. Σας παρακαλώ ένα λεπτό. Γιατί δεν είναι τελευταία φορά που το συζητάμε, μόνο η πρώτη φορά. Ακόμη δεν είχαμε καν την έκθεση του κύριου Νόιζερ. Ευχαριστώ. Η ερώτηση του κυρίου Φιέλνερ. Πόσο έχει συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών. Ναι, συμμετείχε. Περισσότερο ίσως από ό,τι σε άλλες περιοχές. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σόου λοιπόν Φυσικά υπάρχει διαφορά μεταξύ συμμετοχής και επίτευξης των ετοιμάτων σου. Και εδώ βλέπω διαφορετικές απόψεις συζήτηση. Ναι λοιπόν, συμμετείχε η κοινωνία των πολιτών. Ερώτηση του κυρίου Νόιζα τώρα για την ε, ΕΠΑ με το Κάρι Φόρουμ και να το συνδυάσω και με το θέμα σωστών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπήρξε πενταετής ε, μελέτη αντικτύπου για το Κάρι Φόρουμ. Ήταν δύσκολο να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα της ΕΠΑ γιατί συνέπεσε με την εφαρμογή της και η οικονομική κρίση. Αλλά τα στοιχεία που έχουμε για το εμπόριο καταδεικνύουν κάποια θετικά αποτελέσματα για τη δομικανή δημοκρατία συγκεκριμένα για ορισμένα προϊόντα και για κάποιους άλλους εξαγωγείς. Για παράδειγμα αυξήθηκαν οι εξαγωγές ρυζιού παράλληλα όμως. Δεν βλέπουμε να έχει θετική επίπτωση στο εμπόριο εντός της περιοχής του Φόρουμ. Σημαντικός στόχος αυτός του Φόρουμ. Και δεν ξέρουμε αρκετά για το τι επίπτωση είχε στη μείωση της φτώχειας, ε, τις εργασιακές σχέσεις και το περιβάλλον. Αν δούμε τους δείκτες ε, για το περιβάλλον, δεν βλέπουμε αλλαγές. Ίσως δεν έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή, ή δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Δύσκολο λοιπόν να εξαχθούν ε, διδάγματα από το Κάρι Φόρουμ για να είναι πρότυπο για τη Δυτική Αφρική. Αλλά πρέπει να το δούμε. Η πενταετής ε, αποτίμηση, δηλαδή μετά από πενταετία, ε, είναι σημαντική, πρέπει να γίνεται. Για τα στοιχεία. Φυσικά συμφωνώ με την κυρία Καλίνη, υπάρχει αυτή η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που έχει διάφορα στοιχεία για την απώλεια εισοδήματος από τους δασμούς. Είδα τη μελέτη για την Ιγυρία είναι. Υπάρχουν και άλλες χώρες στην περιοχή. Έχουμε την κατάσταση μετά το έμπολα, Γουινέα, Λιβερία. Ποια θα είναι η επίπτωση και στο Μαλί όπου υπάρχουν τόσες πολλές διανέξεις. Δεν έχω δει πρόσφατες μελέτες για τις επιπτώσεις των ΕΠΑ σε αυτές τις χώρες που είναι επίση στην περιοχή αυτή. Έγινε μια άλλη μελέτη για την Κάνα από την ε, υπηρεσία μελετών του Υπουργείου Εξωτερικών της ε, Ολλανδίας η Γκάνα είναι ισχυρή οικονομική δύναμη στην περιοχή αλλά η μελέτη αυτή λέει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει η συμφωνία αυτή σε περισσότερη ανισότητα μεταξύ του βορρά και του νότου της χώρας όλα αυτά νομίζω ότι είναι φανερό ότι μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλες οι μελέτες πρέπει να είναι αναλυτικές και σε βάθος ε, για να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει μια τέτοια συμφωνία στην Κάνα, την Ιγυρία και άλλες χώρες. Για το φορολογικό εισόδημα, ναι, να το δούμε το θέμα προσεκτικά. Ποιε θα είναι οι μειώσεις και ποιε αντισταθμίσεις μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την ανοιχτή πρόσκληση από την κυρία Αγκαλίνα της Επιτροπής να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επιτήρησης. Η κοινωνία των πολιτών ήδη συμμετέχει μέσω της ε, κοινή συμβουλευτική Επιτροπής για το Κάρι Φόρουμ και αν ε, τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία για το ECOWAS βεβαίως η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετάσχει στην ε, παρακολούθηση εφαρμογής. Ε, Πρόεδρο, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει χρόνο, δεν μπορείτε να απαντήσετε όλε τι ερωτήσει. Θα επανέλθουμε για το θέμα αυτό. Υπάρχει κάτι επίγον που θέλετε να πείτε τώρα. Α, θέλετε να ακούσετε το τελευταίο. Καλά, να το ακούσετε. Ωραία, το τελευταίο. Για τα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να περιληφθούν στην μελέτη επιπτώσεων και από ό,τι κατάλαβα αυτά που είπε ο πρόσωπο ΕΚΟΒΑΣ, ε, του ικανοποιεί πλήρω ε, η εξαίρεση που παρέχεται για τα γεωργικά αλλά διαπιστώνω ότι υπάρχουν ακόμα ανησυχίε για το γαλακτοκομικό τομέα, για τη σκόνη γάλακτο. Μα δεν είπα αυτό. Είπα ότι προστατεύεται ο γεωργικό τομέα. Προστατεύεται. Ναι, έτσι το κατάλαβα, λέει ο κύριο Έβερτ. Ναι, ναι, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Νόρμπερτ, θε πάλι το λόγο. Πολύ χρήσιμη συζήτηση και χαίρομαι που την ξεκινήσαμε έγκαιρα Οπότε έχουμε πολύ καιρό, Νόρμπερτ. Γιατί το φθινόπωρο θα υποβάλει την έκθεσή σου. Ευχαριστώ θερμά και τους καλεσμένους μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, μας έχουν απομείνει ελάχιστα λεπτά. Οι διερμηνείς μας έδωσαν και ένα τέταρτο επιπλέον το πολύ για να συζητήσουμε το σημείο 16 για τις κλιματικές αλλαγές και την συνεισφορά μας στην Σύμβαση των Παρισιών. Ώρα των ερωτήσεων αναβάλλετε για την επόμενη σε το σημείο 17 δηλαδή. Και παρακαλώ όσοι φύγουν να το κάνουν αθόρυβα. Και η συνομιλία σας παρακαλώ εκτός αιθούσης. Φύγετε αθόρυβα. Λίγος χρόνος μας έχει μείνει, γι' αυτό θα γίνει μια προκαταρκτική συζήτηση πριν την προθεσμία για τις τροπολογίες και το κυρίως θέμα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου και θα προβλέψουμε περισσότερο χρόνο για πιο εμβριθή συζήτηση. Ε, βάλτε τα ακουστικά σας. Ε, μερικές φορές ε, με το θόρυβο ε, καλύτερα ακούτε με τα ακουστικά από ότι χωρίς. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Οι διερμηνείς μας έδωσαν ακόμη ένα τέταρτο το πολύ. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε κατάχρηση της υπομονής τους. Προτείνω λοιπόν σήμερα να γίνει μια σύντομη συζήτηση πριν την προθεσμία για τις τροπολογίες και στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου θα έχουμε πιο εκτενή ευρυθή συζήτηση αν χρειαστεί. Γιατί το θέμα όντως είναι πολύ σημαντικό και λυπάμαι που πρέπει να το στριμώξουμε στο τέλος της συνεδρίασης. Σύντομη λοιπόν συζήτηση σήμερα. Να ε, επισημάνουμε κάποια σημεία που θέλουμε να τροποποιήσουμε στο ψήφισμα της κυρίας Ζαμπόρσκα και τις λεπτομέρειες θα τις δούμε στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Αποουσιάζει η κυρία Ζαμπόρσκα που είναι η συγγετριά μας, ο κύριος Στίερ θα την αντικαταστήσει. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς η Άννα Ζαμπόρσκα κολλείεται. Μου ζήτησε όμως ε, να διαβάσω τα σχόλιά της ε, για την έκθεση. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω γρήγορα μένα αλλά με τρόπο που να γίνει κατανοητός. Οι προσπάθειες να περιοριστούν, να, να, το, να περιοριστεί το τίμα των κλιματικών αλλαγών είναι σημαντικές. Είναι σημαντική πρόκληση για το περιβάλλον, τη βιομηχανία, το εξωτερικό εμπάριο και τη διπλωματία. η η διάσκεψη των Παρισίων στο Δεκέμβριο του 2015 θα διαδραματίσει ρόλο στις αναπτυξιακές πολιτικές για δύο λόγους. Οι κλιματικές αλλαγές καταρχήν συνιστούν μείζωνα απειλή για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες γιατί έχουν ελάχιστους ή καθόλου, καθόλου πόρους για να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες ε, συνέπειες στο περιβάλλον τους. Πολλές χώρες ε, αντιμετωπίζουν κρίση εξαιτία της λειψιδρία, τη επιδείνωση του εδάφους, αντιμετωπίζουν πείνα και υποσυτισμό. Ενώ σε άλλες χώρες χάνουν ε, γη καλλιεργήσιμη όσο ανεβαίνει το επίπεδο της θάλασσας. Είναι σημαντικές αυτές οι εξελίξεις ε, σε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που έχουν παλιές τεχνολογίες για την, παραγωγή ενέργεια και τροφίμων και σημαντικό αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα. Μάλιστα οι χώρε αυτέ δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τι ε, πεπαλαιωμένε τεχνολογίε του. Θα πρέπει οποιοδήποτε σχέδιο δράση ε, που στόχο έχει τη μείωση τη της του πλανήτη και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των αναπτυσσομένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Γι' αυτό σα καλώ να στηρίξετε τις ε, συστάσεις της γνωμοδότησής μου που ε, επισημαίνουν την τροτότητα του αναπτυσσόμενου κόσμου και το σχετισμό της, ε, των κλιματικών αλλαγών, των μεταναστευτικών ροών και τον κίνδυνο συγκρούσεων για την ε, εκμετάλλευση των πόρων. Θα πρέπει να μειωθούν βέβαια οι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, να μην κλιμακωθεί η κρίση μεταναστευτική στη Μεσόγειο. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού τι ευθύνε του, ανεπτυγμένε και αναπτυσσόμενε χώρε για να υλοποιήσουν του στόχου που θα θεσπιστούν στη διάσκεψη των Παρισίων. Η έκθεση Παρνιέ είναι πολύ φιλόδοξη, ζητά περαιτέρω μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από 40 50, σε 50% μέχρι το 2030. Δεν είναι δικό μα ρόλο ε, να συζητήσουμε κατά πόσο είναι ρεαλιστική ε, η ιδέα σε ένα πλαίσιο ε, υψηλού παγκόσμιου ανταγωνισμού και μια βιομηχανία προσπαθεί να ανανύψει από την ύφεση. Ευθύνη μας είναι να τονίσουμε την ανάγκη διαλόγου με τις αναπτυσσόμενες χώρες και την απαραίτητη συνοχή μεταξύ των κλιματικών στόχων και των αναπτυξιακών μας προσπαθειών. Και γι' αυτό προσβλέπω σε περαιτέρω αγαστή συνεργασία επί της γνωμοδότησής μου. Αυτά λέει η κυρία Ζαμπόρσκα στο κείμενο που σας διάβασα. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό που είπα και στην αρχή. Δεν πρόκειται να τροποποιήσουμε εμείς τους στόχους ε, για τη μείωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ε, παρακάλεσε να περιοριστούμε σε ένα σαφές μήνυμα, γιατί πέρυσι είχαμε πληθώρα τροπολογιών και καμία δεν πέρασε γιατί ήταν μεγάλος ο αριθμός τους. Ας προσπαθήσουμε φέτος να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα θέματα, να εστιαστούμε σε δικές μας προτεραιότητες και έτσι θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να ασκήσουμε κάποια επιρροή, να έχει βάρος και η δική μας γνώμη. Βέβαια δεν ήμασταν όλοι πέρυσι, μερικοί είμαστε καινούργοι και δεν... γι' αυτό το λέω για να καταλάβουμε πώς λειτουργούμε. Ο Τζέιμς πρώτα και μετά η Μαρία. Ο Σεπ ο πρώτος που είναι ο σκιώδης ηγητής για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της και τον κύριο Στίρ για την ε, αντικατάσταση και την παρουσίαση της γνώμης της. Θα είμαι λακωνικός. Θα ήθελα να πω ότι όταν μιλούμε για τις κλιματικές αλλαγές και την επικείμενη διάσκεψη κορυφής των Παρισίων, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η ανάπτυξη να μην γίνει ένα επιπλέον θέμα, ένα παρεμπίπτον θέμα που θα στριμωχθεί στο τέλος. Να γίνει ένα απόσπαστο τμήμα η ανάπτυξη όλων των διεθνών αναπτυξιακών μας στόχων. Γνωρίζουμε ότι οι κλιματικές αλλαγές και η ανάπτυξη είναι η διόψη του ίδιου νομίσματος και η πρόοδος στη συζήτηση για τη συνέπειες των κλιματικών αλλαγών περιλαμβάνει και τη συζήτηση για την απειλή στα οικοσυστήματα και τον τρόπο που επηρεάζεται η ζωή όλων των κατοίκων του πλανήτη και ιδιαίτερα εκείνων που διαμένουν στις πιο ευάλωτες και φτωχότερες περιοχές του κόσμου που είναι και πιο τρωτοί και ευάλωτοι απέναντι στις κλιματικές αλλαγές. επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, αλλά και στη Βόρεια Αμερική και σε άλλες περιοχές του κόσμου και σε πιο ανεπτυγμένες χώρες. Έχουμε, οι χώρες αυτές έχουν αναπτυχθεί κυρίως με ορυκτά καύσιμα. Οι χώρες αυτές έχουν ιδιαίτερη ευθύνη και θα πρέπει να μεριμνήσουν στο μέλλον η ανάπτυξη να μην γίνει εις βάρος του πλανήτη και να μην πληρώσει το τίμημα της ρήπαση του πλανήτη, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να δίνουμε εμεί μαθήματα για βιώσιμη ανάπτυξη, όταν εμεί οι ίδιοι ε, ιστορικά έχουμε θετήσει διαφορετική πορεία. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και να ενθαρρύνουμε μετά τις αναπτυσσόμενες χώρες να κάνουν το ίδιο. Και υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας. Θα πρέπει να τονίσουμε στην δική μας γνωμοδότηση ότι προβλήματα που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές, έλλειψη πρόσβασης στο είδωρ, στις αρρώσιμες αιγαίες, δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας στις αναπτυσσόμενες χώρες με μακροπρόθεσμες συνέπειες και σε εμά. Την περασμένη εβδομάδα κάποιος από το τσάντ μας είπε ότι αν κάποιος δεν μπορεί να παράγει τρόφιμα για την οικογένεια, φυσικά ε, θα υποκύψει στις ε, σιρήνες εκείνων που προσφέρουν ε, ευημερία. Κάτι που θα δημιουργήσει αστάθεια. Χαίρομαι που αναγνωρίζουμε τη μείζωνα απειλή που συνιστά κάτι τέτοιο για τις αναπτυσσόμενες και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Το θέμα αυτό θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για τις κλιματικές αλλαγές και να θεωρήσουμε και το μεταναστευτικό κύμα στη Μεσόγειο ως πρόβλημα ε, που σχετίζεται και με τις κλιματικές αλλαγές. Ε, δεν είναι όμως μόνο περιβαλλοντικό το πρόβλημα, είναι και κοινωνικό και αναπτυξιακό. Γι' αυτό και η γνωμοδότηση έχει μεγάλη σημασία. Η κυρία Χόιλμπορ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ για αυτή την έκθεση της κυρία Ζαμπόρσκα, διότι νομίζω ότι η έκθεση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή, περιέχει πολύ σημαντικά στοιχεία για τους ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους τους θέτει στο επίκεντρο και τονίζει ότι δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τους στόχους αυτούς της ανάπτυξης μη επιτυχάνοντας ε, να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς και τη σχέση με τους πρόσφυγες και τις μεταναστευτικές ροές μπορούμε να την αναπτύξουμε λίγο αλλά αναφέρεται μία πλευρά που δεν περιέχεται και που νομίζω ότι είναι σημαντική πλευρά για μας είναι ότι είναι μοναδική ευκαιρία για να συνδέσουμε την αλλαγή του κλίματος με την εργασία των ΗΕ για το θεματολόγιο μετά το 2015 είναι ένα θέμα που συνδέεται με την αναπτυξιακή πολιτική θα έπρεπε να τονιστεί σε αυτήν την έκθεση. Το άλλο σημαντικό είναι πώς θα χρηματοδοτήσουμε την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει αυτό να είναι στο κέντρο της διάσκεψη στο Παρίσι, γιατί αν δεν υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση, οι αναπτυσσόμενε χώρε δεν θα τηρήσουν τι υποχρεώσει του. Δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τα μέτρα προσαρμογή. Πρέπει ω Επιτροπή Ανάπτυξη να ε, τονίσουμε αυτή τη σύνδεση. Και τελευταίο σημαντικό σημείο είναι η αναπτυξιακή συνεργασία. Πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο τις αναπτυσσόμενες χώρες για βιώσιμη γεωργία, που θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Οι χώρες αυτές και η γεωργία τους, οι γεωργοί τους είναι οι πρώτοι που θίγονται και αυτοί που θίγονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να αναφερθεί και αυτό. Και η μικρή κλίμακα γεωργία πρέπει να υποστηριχθεί και να υπάρξει διαφοροποίηση των καλλιεργειών σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον και οικολογικές ε, καλλιέργειες να στραφούμε. Είναι σημαντική σύνδεση μεταξύ αλλαγής του κλίματος και ανεπτυξιακής συνεργασίας. Και θα αποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε περισσότερο στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Δεν ε, είδα να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Η κυρία Μπάντρα από τη Γενική Διεύθυνση Κλίν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Θα επιχειρήσω να είμαι πολύ σύντομη. Καταλαβαίνω ότι είμαστε υποπίεση χρόνου. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την γνώμη της, τη γνωμοδότηση που θα κάνει. Τα σημεία που αναφέρθηκαν στη γνωμοδότηση δείχνουν καλή κατανόηση των διακύβευμάτων. Η προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη ε, σαφώς επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, τις ξηρασίες λοιπόν, ε, να σταθεί και μη προβλέψιμο καιρό. Όλα αυτά οξύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν και λόγω των ανισοτήτων. Η συνδιάσκεψη COP21 στο Παρίσι θα είναι σημαντική ευκαιρία για να ξεκινήσει μια επιτάχυνση προς την οικονομία χαμηλής εκπομπής άνθρακα. Γιατί θα ισχύει για όλες τις χώρες ή οποιαδήποτε συμφωνία. Δεν θα υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ε, διαχύσεις αρμοδιότητας με βάση την κατηγορία χωρών που είχαμε από το 92, την κατηγοριοποίηση δηλαδή χωρών. Θα υπάρχει δηλαδή εφαρμογή παντού από όλες τις χώρες των αρχών της ε, Σύμβασης των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή. Και έτσι θα αντιμετωπίσουμε πιο στεναρά τα προβλήματα. Είναι σημαντικό αυτό. Και η αναπτυξιακή συνεργασία είναι μία από τις πολύ βασικές πτυχές της ε, διπλωματίας για το κλίμα. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες συνεργασίας, τις δυνατότητες ε, κοινής δράσης για να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή και την ε, ανεπτυξιακή συνεργασία. Οι αναπτυσσόμενες χώρες παράγουν το 75% των εκπομπών σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι πιο ευάλωτες χώρες, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, είναι αυτές που έχουν ε, τις λιγότερες δυνατότητε να δράσουν και αντιμετωπίζουν δυσανάλογες ε, απαιτήσει. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να τις στηρίξουμε με διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Η γνωμοδότηση τονίζει τη δέσμευση της Ένωσης και άλλων αναπτυγμένων χωρών για τα 100 δις. Εδώ χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη, καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική. Γιατί πολλές φορές ε, ακόμη και τα νούμερα παραποιούνται όπως παρουσιάζονται. Καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το τονίσει αυτό. Όχι μόνο για το θέμα της χρηματοδότησης, αλλά και για το θέμα της ε, διαφάνειας των μέτρων μείωσης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δεν στηρίζουμε ένα στις προσπάθειε του άλλου. Δεν έχουμε λοιπόν πολυμερή εφαρμογή ουσιαστική. Η διαφάνεια, η δημιουργία εμπιστοσύνη, η κατάδειξη του ότι εφαρμόζουμε τι δεσμεύσει μα, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να μπουν στο σχέδιο γνωμοδότηση. Δεν ξέρω αν η συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση Ντεύκο, θέλει να προσθέσει. Ευχαριστώ. Είμαι η Χριστιανά Καύσκα Πάλμερ ε, και ευχαριστώ την Επιτροπή και την Πρόεδρο που μας καλέσατε να είμαστε σήμερα εδώ. Ίσως για να συνεχίσω με βάση τα όσα είπατε για τη χρηματοδότηση. Το τμήμα της χρηματοδότησης βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης και από την πλευρά μας πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε Μία εκτίμηση 40 δις ευρώ ανάμεσα στο 2007 και το 2020 θα αφιερωθούν σε δραστηριότητες σε σχέση με το κλίμα μέσω των διαφόρων εξωτερικών μέσων. Δύο δις ετησίως δηλαδή είναι μεγάλο ποσό νομίζω και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού θα πάει στις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, γιατί αυτές είναι που φέρουν το μεγαλύτερο κόστος των κλιματικών αλλαγών ε, δεν μπορούμε λοιπόν να χωρίσουμε την ανάπτυξη από τις κλιματικές αλλαγές. Είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Το ίδιο σημαντικό, πέρα από την άμεση αυτή συνεισφορά, είναι η ιδέα της ε, ε, καινοτόμας χρηματοδότησης ε, ε, ως έναν τρόπο να μοχλεύσουμε και να αυξήσουμε τον αντίκτυπο των, ε, της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Από το 2007 πάνω από 1,2 δις ε, ε, ε, χρηματοδότησης κινητοποίησαν ακόμα 25 δις και, ελπίζουμε, και, και υπολογίζουμε ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο αυτός ο αριθμός. Και κάτι για τη γεωργία και το γεγονός ότι επίσης εστιάζουμε στο mainstreaming του περιβάλλοντος και των κλιματικών αλλαγών στους τομείς κλειδιά όπως η γεωργία, όπου η σχέση ανάμεσα στο κλίμα και τη γεωργία είναι φυσικά ε, στόχος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι η υποβολή προθεσμιών ε, θα γίνεται μέχρι τις 2 Ιουλίου και θα ψηφίσουμε στη συνεδρίασή μας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές που θα είναι στις 3 Σεπτεμβρίου και όχι την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Γιατί πολλοί συνάδελφοι έλεγαν ότι δεν είναι καλύτερη ιδέα να ψηφίσουμε την πρώτη Δευτέρα μετά τι διακοπέ. Δεν έχω δει τίποτα να έχει ζητήσει κανείς για τα διάφορα. Να ευχαριστήσω ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους Δερμηνείς. Είχαμε μια μεγάλη μέρα, μακριά μέρα και εσείς με βοηθήσατε και είχαμε και πολύ γρήγορους ομιλητές σήμερα. Ξέρω λοιπόν πως ε, πολύ δουλέψατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε και πάλι και εμείς σας ευχαριστούμε οι Δερμηνείς. 13 Ιουλίου η συνεδρίαση έχει ακυρωθεί. Σας ευχαριστώ. Yeah, thank you. We, it was an opportunity to do some quiet work.